Okay, friends and... Αγαπητοί φίλοι και προσκεκλημένοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε μια ελαφρά καθυστέρηση. Ελπίζω ότι θα έχουμε και μέλη του Κοινοβουλίου που θα έρθουν όταν θα έχουν χρόνο και ίσως θα φύγουν και θα ξανάρθουν. Ε, Γιατί είναι μια σημαντική συνεδρίαση αυτή για μας ώστε να ακούσουμε τους νέους, όχι μόνο στις οικογένειές μας, αλλά και από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Να ακούσουμε τι σκέφτονται οι νέοι για το μέλλον τους, το δικό μας μέλλον. Και πώς ε, θέλουν να καταλήξουν ε, στη ζωή αλλά και στην εργασία. σε μια κατάσταση να σκέφτεσαι ε, ότι είσαι ικανοποιημένο από τον εαυτό σου και να αποκτήσει κάτι για το οποίο αγωνίστηκε. Αυτή είναι η τρίτη ε, εκδοχή της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για την Νεολαία που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο στις αρχές Ιουνίου 2018. Και σήμερα έχουμε το follow-up, τη συνέχιση σε αυτή την ε, τρίτη Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεονέα. Περίπου 9.000 ε, νέοι συζήτησαν κατά την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεολαία στο Στρασβούργο ιδέες και προτάσεις για την Ευρώπη το αύριο. Και με αυτό ασχολούμαστε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Γενοβούλιο Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, πώς θα αναπτυχθεί η Ευρώπη, πώς θα εξελιχθεί. και τι σχεδιάζουμε για την Ευρώπη του αύριο. This, ε, youth Αυτή η ακρόαση για την νεολαία ε, οργανώνεται προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα καλό follow-up ε, της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για την νεολαία και έχω την χαρά να καλωσορίσω τρεις νέους συμμετέχοντες που παρευρίσκονται στη συνεδρίασή μας για να μας παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε θέματα που σχετίζονται με τα θέματα της Επιτροπής μας. Εξιότητες για τις ε, μελλοντικέ θέσεις εργασίας και είσοδος στην επασχόληση. Το μορφότυπο της εκκρόασής μας το καλούμε έλεγχο ιδεών, ideas check. Είναι ένα ειδικό μορφότυπο που έχει αναπτυχθεί για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεολαία. Οι τρεις νεαροί θα μας δώσουν τις ιδέες τους και εμείς ως μέλη του Κοινοβουλίου θα είμαστε αυτοί που θα συλλάβουν τις ιδέες θα αναπτύξουμε και θα συζητήσουμε τις ε, ιδέες που θα παρουσιαστούν σε αυτό το μορφότυπο. Να παρουσιάσω τους ομιλητές. Καταρχήν ο Άρθρου Κοράτσα από την Αυστρία. Θα μας παρουσιάσει τις ιδέες του για μια χάρτα του εργατικού δυναμικού διαγενειακού χαρακτήρα και για περισσότερη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο Erasmus η Γκίλμετ Ντεζάν από τη Γαλλία θα παρουσιάσει ιδέες για μια πλατφόρμα για εξειδικευμένους πρόσφυγες για να καλύψουν ρόλους στον τομέα της εκπαίδευσης και ιδέες για ένα κολαπτήριο επιχειρήσεων, ένα πρόγραμμα κολαπτήριου επιχειρήσεων για τους πρόσφυγες. Και ο Κρίστιαν Μόλμπι από τη Δανία θα μας παρουσιάσει ιδέες για την επιχειρηματική εκπαίδευση και για τις μαθητείες ε, κατά τη διάρκεια του σχολείου. Δεν πρόκειται λοιπόν για φαντασίες εδώ, πρόκειται για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ιδέες για το μέλλον. Και φυσικά αυτά θέλουμε να συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή. Θα σας ε, δώσω 3-4 λεπτά στη διάθεσή σας. Τέσσερα δεν είμαι τόσο αυστηρή. Και κατόπιν το λόγο θα έχουν οι βουλευτές για να αντιδράσουν. Ε, ε, και κατόπιν θα θέσουμε ερωτήσεις στους προσκεκλισμένους μας και θα προβούμε στη συζήτηση. Θα ξεκινήσω δίνοντας το λόγο σε σένα, Άρθουρ. Προσπάθησα να μην ακρηγορήσεις. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα. Η πρώτη ιδέα από την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεολαία που σας παρουσιάζω αφορά το θέμα της απασχολησιμότητας και της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων. Ο χάρτης ε, που θέλω να παρουσιάσω προσπαθεί να ενθαρρύνει τις οργανώσεις να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο χώρο εργασίας ε, που να οδηγεί σε μεταφορές δεξιοτήτων. Αυτό θα υποστηρίξει ε, την διαβίωμάθηση, το πρώτο αρχή στον πυλώνα των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Εγώ, καθώς είμαι ε, στην ηλικία των 20, είναι λογικό ότι βλέπω τον εαυτό μου να αλλάζω δουλειές στο μέλλον και ίσως να επιστρέφω και στο σπίτι που μεγάλωσα. Μία πτυχή της πραγματικότητας των νέων σε αυτόν τον κόσμο που γρήγορα αλλάζει είναι η πρόκληση να οικοδομήσουν ε, σχέσεις μακροπρόθεσμες ε, στο χώρο εργασίας και τα διαγενειακά θέματα ε, για να ε, θα βοηθήσουν τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες. Αυτές οι σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μεταφορές δεξιοτήτων προκειμένου να απαντηθούν κάποιες ελλείψεις όπως η έλλειψη δεξιοτήτων βασικών των νεαρών εργαζομένων και χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες του μεγαλύτερου σε ηλικία προσωπικού. Χρειαζόμαστε πραγματική για να ενδυναμώσουμε τους κοινωνικούς δεσμούς. Αυτός ο διαγενειακός χάρτης θα είναι ένας εθελοντικός κώδικας πρακτικής που θα ορίζει ένα σύνολο ε, προτύπων. Αυτά τα πρότυπα θα σκοπεύουν να ενδυναμώσουν ε, την κουλτούρα της μάθησης της οργανώσεις και να υποστηρίξουν διαγενειακές μεταφορές δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα πρότυπα θα απαιτούσαν μια διαγενειακή ισορροπία στην ε, στο εργατικό δυναμικό, ε, σχέσεις καθοδήγησης μεταξύ νεαρών και έπειρων εργαζομένων ε, και μια ποιότητα καθοδήγησης. Αν μια εταιρεία αποφασίσει να δεσμευτεί με τα πρότυπα αυτά, θα μπορούσε να κάνει αίτηση στο, στον αντίστοιχο εθνικό οργανισμό που είναι αρμόδιος για το Erasmus Plus ε, και να αποκτήσει μια επίσημη πιστοποίηση. κατόπιν, μια διαδικασία παρακολούθησης θα μπορούσε να διασφαλίσει την ποιότητα της δέσμευσης καθοδήγησης αυτή η διαπίστευση ε, θα μπορούσε να δηλώνει την ποιότητα ε, των χωρών εργασίας όσων ζητούν δουλειά και να δίνει σε εταιρείε ε, ένα προβάδισμα ε, στην πρόσληψη και στην διατήρηση του προσωπικού επίσης. Οι εταιρείε θα μπορούσαν να αποκτήσουν μια καλύτερη φήμη για κοινωνική ευαισθητοποίηση και να προωθήσουν τη χάρτα σε οργανώσει που δεν έχουν αποκτήσει διαπίστευση. Αυτός ο Ευρωπαϊκός Χάρτης θα κεφαλοποιούσε διάφορες διαγενειακέ δεξιότητε δραστηριότητε επίση θα δημιουργούσε μια κουλτούρα που θα υποστήριζε περισσότερο του κοινωνικού δεσμού και τη διαβίου μάθηση. Έτσι λοιπόν, σα απευθύνω έκκληση να θεσπίσετε ένα διαγενικό χάρτη για το εργατικό δυναμικό. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην ε, κυρία ε, ε, Ζούλια Μινιέτ. Κυρία Μουρανσόρφη, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για να συλλέξουμε λοιπόν αυτές τις ιδέες θα πρέπει να επεξεργαστούμε την παρουσίαση που ακούσαμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση. για αυτό το χάρτη της εργασίας ε, μεταξύ των γενεών και την σφραγίδα αυτή που υπάρχει στις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Η πρώτη ερώτηση. Γνωρίζουμε ότι όπου μιλάμε για εκμάθηση, η ποιότητα προφανώς ε, του ατόμου, του μέντορα που δίνει την κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχετε κοιτάξει το θέμα του πιστοποιητικού ποιότητα σε ό,τι αφορά τον ε, δάσκαλο, τον, ε, το άτομο που δίνει την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Δεύτερη ερώτηση. Μιλήσατε για δεξιότητες, για προσόντα και διαπιστώσατε ότι στα στην επαγγελματική σας ζωή θα γνωρίσετε όλο και πιο πολλά επαγγέλματα, με αυξανόμενο χαρακτήρα. Αλλά περνάμε από την ε, διάσταση των προσόντων σε διάσταση των ικανοτήτων. Αυτές οι ικανότητες λοιπόν που μεταφέρονται από δουλειά σε δουλειά, αυτές είναι που επιτρέπουν στους νέους να μην κινούνται μόνο σε μία σταδιοδρομία, αλλά μπορούν, να μπορέσουν να αλλάξουν δρόμο. Αυτές είναι λοιπόν οι δύο που ήθελα να σας θέσω για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. very for your questions. Um, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά τώρα το πρώτο, όσον αφορά την ποιότητα των μεντόρων, Φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ελέγχου ε, σχετικά με το πώς ορίζουμε την ε, ποιότητα ε, του μέντορα, πώς ορίζουμε ακριβώς την ποιότητα. Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα και το πώς θα παρακολουθείτε επίσης. Μία εναλλακτική λοιπόν θα ήταν να αξιολογείται με υποκειμενικό τρόπο, δηλαδή να υποβάλλονται έρευνες, ε, μελέτες, ε, ερωτηματολόγια από συμμετόχοντες οι οποίοι θα εκτιμούν ε, την ικανοποίησή τους. Η έμφαση λοιπόν δίνεται σε μια διαδικασία, διαδικασία μάθησης και από τις δύο πλευρές ε, όπου οι νέοι θα αποκτούν ε, ψηφιακές δεξιότητες και άλλες και είναι σημαντικό λοιπόν και οι δύο πλευρές ε, αυτής της με τουρκικές σχέσεις να μπορούν να εκφράσουν την ικανοποίησή τους. Αυτό είναι ένας τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας. Άλλα τώρα μέσα θα μπορούσαν να επικεντρώνονται στο ίδιο το μαθησιακό αποτέλεσμα ή σε άλλα μέτρα όπως είναι για παράδειγμα το ε, αποτέλεσμα της ε, εργασίας. Τώρα όσον αφορά την επαγγελματική κινητικότητα και το δεύτερο σας ερώτημα θεωρώ ότι είναι μια βασική προσέγγιση για τη συγκεκριμένη ιδέα που εφοπλίζει τους νέους ε, με δεξιότητες που θα μπορέσουν να τους κάνουν να κινηθούν καλύτερα στον εργασιακό χώρο. Υπάρχει μια έκθεση από την ΣΕΝΤΕΦΟΠ που τονίζει το θέμα της ε, ε, μη σωστής αντιστοίχησης των δεξιοτήτων και ε, υπάρχουν σε αυτό το θέμα το αίσθημα της, ε, του πολίτη, η προσαρμοστικότητα και αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούν να συμπεριλαμβάνονται, οπότε θεωρώ ότι ενισχύοντας τους κοινωνικούς δεσμούς με πιο έμπειρους εργαζομένους, οι νέοι θα μπορέσουν να κερδίσουν και αυτό το πολιτιστικό κεφάλαιο, το οποίο ε, παθητικά κληρονομείται και δεν μαθαίνεται ενεργητικά στην σύγχρονη ε, παιδεία. Ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να σας απάντησα στο ερώτημά σας. Ωραία. Θα επανέλθουμε σε εσά, όμως για την ώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Γκουιμέτ ε, Τεζόν. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Ξέχασα. Το ξεχνάμε μερικές φορές στο Κοινοβούλιο. Όμως έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οπότε θα ήθελα αρχικά να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, πρόσκληση. Όσο γνωρίζετε, η Επιτροπή είναι, ε, επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε δράσεις που αφορούν νέους και χαιρόμαστε να μαθαίνουμε ιδέες ε, για το μέλλον και ήταν ε, σημαντικό για μένα το να ακούσω στην εισαγωγή του άρθρου του Άρθουρ την αναφορά στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα. Νιώθω πιο ήρεμη έτσι. Όταν το υιοθετούν αυτό οι νέοι, όταν ξέρουν περί τίνος πρόκειται και προσπαθούν να αναπτύξουν ιδέες που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο πυλώνα, τότε πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας ένα φωτεινό μέλλον. Εκτιμώ επίσης την ιδέα ε, αυτού του ε, χάρτη ε, που πραγματικά θα αποτελήσει μια πρόκληση για το δημογραφικό μας μέλλον. Αυτές οι διαγενειακές σχέσεις αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο της δικής μας πολιτικής κατάρτισης διότι θεωρούμε ότι αυτό το οποίο θέσαμε ως βάση το 2011 στην ε, ημερήσια διάταξη για την ενήλικη μάθηση που αφορά την ενίσχυση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης για τους ενήλικες μεταξύ των οποίων και ο θελοντισμός και η ε, διαγενειακή μάθηση ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες των ηλικιωμένων για, την, για όφελος ολόκληρης της κοινωνίας είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει ιδιαίτερο σε μια τέτοια χάρτα. Επίσης η πρωτοβουλία αυτή ακολουθήθηκε από το Ευρωπαϊκό Έτος για την ε, διαγενειακή επικοινωνία και τόνισε τις δυνατότητες και ευκαιρίες χρήσης ε, γνώσης που έχει ήδη αποκοντηθεί για να βοηθηθούν οι νέοι, ούτως ώστε πιο γρήγορα και πιο εύκολα να βελτιωθούν και να βρουν εργασία. Πιστεύω λοιπόν ότι η διαγενειακή μάθηση αποτελεί το βασικό στοιχείο του οράματός μας και είμαστε έτοιμοι να δούμε το πώς θα υλοποιηθεί αυτό μελλοντικά. Τώρα, όσον αφορά τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, υπάρχουν αρκετές αρχές οι οποίες συνεισφέρουν προς ε, αυτή την ιδέα. Ε, το δικαίωμα στην συνεχιζόμενη μάθηση, την ίσομη αντιμετώπιση όσον αφορά την απασχόληση και την ε, παιδεία όσον αφορά τους μισθούς, και θα ήθελα επίσης να σας ε, θυμίσω κάποιες συζητήσεις που γίνονται αυτές τις ημέρες της διαπραγματεύσεις όσον αφορά την ε, οδηγία για την ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ε, ζωής που εισάγει το δικαίωμα των γονέων να πάρουν άδεια για να φροντίσουν τα παιδιά τους και να γίνει πιο ισότιμα η κατανομή των ευθυνών και να προσφερθεί και περισσότερη ευελιξία ε, στην εργασιακή ζωή και επίσης να ε, βοηθήσουμε στο γενιακό πλαίσιο. Θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμα ένα πρόγραμμα Κούντβι το οποίο αποτελεί εργαλείο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διανομή γνώσης μεταξύ νέων και ηλικιωμένων και σε αυτό δίνεται η δυνατότητα σε συνδιοξιδοτημένους να λειτουργήσουν ως μέντορες για νεότερους ε, ανθρώπους και να μπορέσουν έτσι να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας. Και επίσης ε, ε, φέρνουμε μαζί μειονεκτούντες ομάδες, ηλικιωμένους και νεότερους για να συνεργαστούν και θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί μια πολύ καλή αρχή της συζήτησης για μελλοντικέ ιδέες καθώς επίσης και μια διατομεακή και διαγενειακή προσέγγιση για την μελλοντική εξέλιξη στην Ευρώπη και ε, χαιρετώ τους νέους για τον ενθουσιασμό τους και την διάθεσή τους να μοιραστούν ιδέες ε, για το τι μπορούμε να κάνουμε μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάκιντάιρ, ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι οι ιδέες σας είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Μου θυμίσατε και ένα πρακτικό παράδειγμα το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται. Και έτσι αυξάνεται η ηλικία του εργατικού δυναμικού στα 10. Και ίσως όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην επιθυμούν ιδιαίτερα να μείνουν στην αγορά εργασία σας. Έχω λοιπόν μια εταιρεία στην περιφέρειά μου, μια εταιρεία μηχανικών που δυσκολευόταν ε, να βρει νέους ανθρώπους να προσλάβει και είχε και εργατικό δυναμικό το οποίο σε ηλικία αυξάνεται. Εισήγαγαν λοιπόν ένα πρόγραμμα μαθητείας και κάθε ένας από αυτούς ε, τους εκπαιδευόμενους είχε ένα μέντορα, έναν από τους ε, πιο ηλικιωμένους εργαζομένους με τρομερή εμπειρία πέρα από τα μαθήματα που έκανε στην τάξη. Αυτό λοιπόν ήταν ε, πραγματικά μεγάλο κέρδο για του νέου που έμαθαν προφανώ πάρα πολλά πράγματα αλλά βοήθησαν και τους πιο ηλικιωμένους γιατί τους έδωσε ένα σκοπό στην επαγγελματική του ζωή. Δεν περίμεναν πλέον ε, την ώρα να βγουν στη σύνταξη. Καταλάβαιναν πόσο σημαντικά ήταν τα προσόντα αυτά που είχαν να μεταφέρουν στου νέους ε, εργαζόμενους. Άρα συνολικά η εταιρεία προχώρησε πολύ γιατί ξαφνικά οι πιο ηλικιωμένοι βρήκαν λόγο ύπαρξη στη ζωή τους, στην επαγγελματική τους ζωή, γιατί επένδυσαν στο μέλλον των νεαρών και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία αυτή και το πείραμα αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Μαρτά έχει το λόγο. Oui. Pardon. Mm, ναι, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Είναι πραγματικά εξαιρετική ιδέα. Γιατί άλλωστε ο πρώτος το στόχος που θα πρέπει να έχετε είναι να μπει ένα αυτή τη μοιραία φράση που διαρκώς ακούν οι νέοι ότι α, δεν έχετε εμπειρία. Θα πρέπει λοιπόν να αποδείξετε ότι είστε διτεθειμένοι να εργαστείτε και αν σας δώσουν την ευκαιρία για να αποκτήσετε την εμπειρία έχετε σκοπό να δουλέψετε και όπως είπατε αυτό ωφελεί και τις δύο πλευρές. Γιατί προφανώς αυτό ωφελεί και τους νέους και τους ε, πιο έμπειρους, τους πιο ολικιεμένους Κάποιες χώρες λοιπόν έχουν προωθήσει τέτοιες ε, πρωτοβουλίες. Στην Ισπανία για παράδειγμα παλιά υπήρχε μια σύμβαση εκπαίδευσης. Αν ήταν λοιπόν μεγάλη ηλικία ή μέση ηλικία σε μία, σε μία επιχείρηση, υπήρχε ένα τέτοιο μέτρο για να εκπαιδεύονται οι νέοι. Γιατί, γιατί και στη βιομηχανία και αλλού σήμερα είναι πολλά ε, επαγγέλματα τα οποία δεν μπορεί να τα μάθει κανείς ε, στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, στη σχολή. Χρειάζονται να τα μάθει κανείς επί τόπου στη δουλειά και έτσι πολλοί, όπως είπε η συνάδελφος, ε, οι ηλικιωμένοι παράλληλα εργαζόμενοι φεύγουν και παίρνουν μαζί αυτή την τεχνογνωσία. Και τρίτον, θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν γιατί δεν είχαν προλάβει την ανανέωση του πληθυσμού που θα έπρεπε να γίνει. Και δεν είχαν προβλέψει να δημιουργήσουν ε, ε, ένα τέτοιο δίκτυο το οποίο θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι εξαιρετική πρωτοβουλία και προφανώς γι' αυτό χρειάζεται χρηματοδότηση. Το Erasmus, το Erasmus Plus θα πρέπει να χορηγούν πιο πολλά κονδύλια για να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγχαρητήρια πάντως για τις προτάσεις σας και τις πρωτοβουλίες σας. Η Πρόεδρος. Να πω δύο λόγια. Πρωτού περάσουμε Συγγνώμη, λέει η πρόεδρος, να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Λαμπαγιώβα. Ευχαριστώ πρόεδρε και θα είμαι σύντομη. Να αναφερθώ στον Άρτορ. Ευχαριστώ που αναφέρες βασικά στοιχεία. Είπε ότι χρειαζόμαστε ευθύνη, ότι χρειαζόμαστε δέσμευση και από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό κλάδο. Χρειαζόμαστε ένα τρίγωνο, το εκπαιδευτικό σύστημα, τους ε, εργοδότες και τους πολιτικούς ηθήνοντες. Χρειάζονται και τα τρία σκέλη για να λειτουργήσει το σύστημα. Ευχαριστώ επίσης που αναφέρατε τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Σε διάφορες περιπτώσεις έχουμε πολλά καλά πραγματά σε επίπεδο κρατών μελών. Αλλά δεν χρησιμοποιούμε επαρκώς αυτή την εμπειρία. Τρίτο θέμα. Ε, η μαθητεία. Αυτό λείπει στην Ευρώπη. Στην ε, Αμερική υπάρχει μεγαλύτερη παράδοση και θα πρέπει να το προωθήσουμε και στα κράτη-μέλη. Τέταρτο σημείο, και εδώ έχω και μια ερώτηση να σας θέσω. Όλοι ξέρουμε ότι ένας καλός συνδυασμό ε, σωστών προσόντων για το μέλλον είναι ένα αμάλγαμα και τεχνικών και πληροφοριακών προσόντων αλλά και πιο ήπιων προσόντων. Η γενιά των 55 και άνω δεν έχει ενδεχομένως ε, τι ικανότητε και τα προσόντα που χρειάζονται στον τομέα τη πληροφορική εσά, τι θεωρείτε ότι σα λείπει πιο πολύ στη δική σα γενιά, μήπως λείπουν ε, τα ήπια αυτά προσόντα και τι θεωρείτε ότι μπορείτε να διδαχθείτε από τι παλιότερε γενιέ. Ευχαριστώ πολύ. Άρθρο, τώρα είναι η σειρά σου, λέει η um, Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με την πρώτη σας ερώτηση. Με τα ποια είδη δεξιοτήτων έχουν νόημα. Αν μιλάμε για τη γενιά Z που είναι η νεότερη γενιά που μπαίνει τώρα στην αγορά εργασίας. Τονίζεται πάντοτε ότι οι βασικές δεξιότητες όπως τα soft skills συγκεκριμένα είναι πολύ σημαντικές και πολύ συχνά λείπουν. Και αυτό σχετίζεται με την όλη συζήτηση για την κοινωνική κινητικότητα και το πολιτιστικό κεφάλαιο που ανέφερα πριν είναι ουσιαστικά μια ενσωματωμένη μορφή συμπεριφοράς και αυτοπαρουσίασης που είναι ζωτική στη σημερινή ώρα εργασίας καθώς οι νέοι συχνά ε, είναι μεμονωμένα άτομα και όχι συλλογική ομάδα που μπορούν να υποστηρίξουν ένα στον άλλο. Και εξού, μάλλον από εκεί ξεκινάει και η ιδέα μου για την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των νέων και των ανθρώπων που μπορούν να τους βοηθήσουν. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για soft skills και βασικές δεξιότητες στην Αυστρία, στην πατρίδα μου. Ένα μεγάλο ζήτημα τώρα είναι η έλλειψη διαθέσιμων μαθητιών σε εταιρείε που αναζητούν μαθητευόμενους για να τους προσλάβουν όμως υπάρχουν ε, περισσότεροι άνθρωποι που ψάχνουν για μαθητείες από τις διαθέσιμες θέσεις τον Ιανουάριο του 2018 είχαμε χίλιες περισσότερες θέσεις από τους ανθρώπους που τις ε, επιζητούσαν και η αιτία θεωρείται ότι ήταν η έλλειψη βασικών αρμοδιοτήτων. Συχνά αναμένεται να έχει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και μια ολιστική εικόνα των δεξιοτήτων των νέων όταν ε, μιλάμε για την είσοδο στην αγορά εργασία. Έτσι λοιπόν αναμένεται να υπάρχουν εμπειρίε ε, σε διάφορους τομεί οι άνθρωποι να παρουσιάσουν ε, διάφορα προσόντα με τις εμπειρίε τους. Αν όμως ο εργοδότης ήξερε ότι ο νέος έχει την δυνατότητα να αποκτήσει στο χώρο εργασίας αυτά τα προσόντα που του λείπουν, μέσω της καθοδήγησης ε, ίσως αυτό θα βοηθούσε και θα ενδυνάμωνε και την ιδέα ότι ο χώρος εργασίας είναι ένας χώρος όπου εξακολουθούν να μαθαίνουν οι νέοι και δεν πρέπει να μπουν εκεί ως ολοκληρωμένα άτομα. Και εγώ νομίζω ότι εδώ επισέρχεται η προσέγγιση που αφορά τα δικαιώματα και μιλάμε για οικονομικούς πόρους όταν η ε, οικονομική διασημότητα των ε, προϋπολογισμών ε, είναι μια συζήτηση που κυριαρχεί. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια αιτήματα από την κοινωνία από τη σκοπιά των δικαιωμάτων ακολουθηθεί κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ για το feedback. Ευχαριστώ. Τώρα είναι η σειρά σας. Έχετε το λόγο, Γκυλμέτ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μας ε, δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε εξ ε, των νέων στην Ευρώπη. Οι ιδέες ε, που θα παρουσιάσω βασίζονται στις ιδέες από την εκδήλωση για την νεολαία και θα χρησιμοποιήσω την πείρα μου. Εργάζομαι ε, στο Chatterbox. Πρόκειται για μια οργάνωση που συνεργάζεται με πρόσφυγες. Η πρώτη μου ιδέα είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την απασχόληση εξειδικευμένων ε, προσφύγων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη. Καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει προσπάθειες στο να συνδέσει τους πρόσφυγες που έχουν προσόντα διδασκαλία με τον κλάδο της παιδείας προκειμένου να ενταχθούν καλύτερα οι πρόσφυγες με προσόντα και να προωθηθεί το εύρος των προσόντων και της εμπειρία των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Αυτός ο μηχανισμός υπάρχει ήδη. Ένα πρόγραμμα που λέγεται Επιστήμη για τους πρόσφυγες έχει ξεκινήσει το 2015 και συντεριά την του ε, που έχουν ιστορικό στις επιστήμες με τα επιστημονικά ιδρύματα είναι προσβάσιμο στους πρόσφυγες και στα ιδρύματα μέσω ε, της πύλης ε, Euraccess. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να διευρυνθεί σε όλο τον κλάδο της παιδείας. θα είναι μια πύλη όπου όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, πανεπιστήμια θα παρέχουν πρόσβαση σε μια σειρά πληροφοριών και υπηρεσίε υποστήριξη σε δάσκαλου πρόσφυγε και εκπαιδευτικού που θέλουν να βρουν εργασία και να συνεχίσουν την σταδιοδρομία του στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει εταιρικέ σχέσει με υφιστάμενε πρωτοβουλίε που ήδη ε, αναφέρουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τους ε, φοιτητές, ε, πρόσφυγες όπως είναι το Refugees Welcome Map ή ε, το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων για τους πρόσφυγες. Τα πανεπιστήμια και τα σχολεία δεν μπορούν να προσλάβουν ανθρώπους χρησιμοποιώντας τους παραδοσιακούς διάβλους, την Chatterbox. Εμείς ε, ουσιαστικά συνδέουμε τους ε, δάσκαλους πρόσφυγες με μαθητές ε, σε όλο τον κόσμο και οι κύριοι πελάτες είναι κορυφαία πανεπιστήμια που αντιμετωπίζουν έλλειψη σε επαγγελματίες των γλωσσών. Πιστεύω ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο ε, από τη δύο πρόσφυγες, ε, τα παιδιά και οι μαθητές ε, που διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που έχουν ιστορικό πρόσφυγα θα ανακαλύπτουν ένα άλλο πολιτισμό, θα ανοίξει το μυαλό τους και θα είναι λιγότερο προκατηλημένοι απέναντι στους πρόσφυγες. Αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017 και ανανεώθηκε φέτος και εφαρμόζεται σε σχολεία στις ΗΠΑ και το ΕΒΑ οι μαθητές είπαν ότι ήταν θετικός ο αντίκτυπος ε, κατά την εισαγωγή ε, ξένων γλωσσών και πολιτισμών στην αίθουσα και αυτό μπορεί να αλλάξει πολλές πόρτες σε οποιαδήποτε σταδιοδρομία και από τη σκοπιά του δασκάλου η έρευνα μου έχει δείξει ότι οι αίθουσε είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για τη μακροπρόθεσμη ένταξη των προσφύγων. Συμπρασματικά πιστεύω ότι η οικονομική και η κοινωνική συμμετοχή καθώς ε, και η προσωπική επιτυχία είναι ζωτική για την αποτελεσματική ένταξη των προσφύγων. Ας δημιουργήσουμε ένα όχημα για την ένταξή τους ε, μέσω ε, μιας απασχόλησης που να έχει νόημα, που υποστηρίζει, θα υποστηρίζει αυτή η πύλη. Και οι πρόσφυγες θα είναι αυτοί που θα βοηθούν, όχι αυτοί που θα ετούνται βοήθειας. Σας ευχαριστώ βοηθούν ε, και δεν ζητούν βοήθεια. Ακούσαμε αντιδράσεις από τους βουλευτές. Θέλει κάποιος να πει κάτι, ο κ. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία. Γιατί πριν 15 μέρε, ε, θυμάμαι ότι ήμουν ε, σε μια γαλλική περιφέρεια, ότι ήρθε να με δει μια καθηγήτρια και μου είπε τι κάνει η Ευρώπη για να αποδεχτεί αυτού του πρόσφυγε. Έχουμε πρόσφυγε με προσόντα. Υπάρχει όμω ε, βέβαια και το πρόβλημα τη αναγνώριση των πτυχίων. Έχετε κάτι κατά νου, γιατί θα πρέπει να βρούμε και μια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Αλλά το κύριο πρόβλημα είναι να μάθει κανεί τη γλώσσα, το είπατε και ε, σίγουρα ε, δεν υπάρχει καλύτερο από το να μάθει κανείς ε, τη γλώσσα. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες κάποιων οργανώσεων, όμως έρχονται απλώ να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν σε εθνικό και κοινωτικό επίπεδο αυτό που προτείνατε μπορεί να μας βοηθήσει να αλλάξουμε την εικόνα που έχει η πλειονότητα για τον πληθυσμό αυτό, γιατί δεν έρχονται εδώ με την ιδέα ότι θα πάρω τη δουλειά κάποιου άλλου ή θα εκμεταλλευτώ από κάποια κοινωνική ε, συνδρομή, όταν δεν έχουν την ε, δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ε, θέλουν να εμπλακούν πλήρως στη ζωή. Σήμερα δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα και όταν κάποιος είναι γιατρός, δικηγόρος, ε, μηχανικός, ε, τεχνικός, δεν σε αποκαλούν ε, πλέον ο μετανάστης ή ο πρόσφυγας, είναι γιατρός, δικηγόρος, ο μηχανικός κτλ. Δηλαδή μιλάμε εδώ για κάποια στοιχεία ένταξης, πολύ ενδιαφέροντα και για αυτούς και για μένα. Στη χώρα μου σήμερα δεν έχουμε γιατρούς και συγκεκριμένα καρδιολόγους. Και δεν υπάρχουν πολιτικές ε, για να βοηθήσουμε αυτούς τους γιατρούς να μάθουν τη γλώσσα και να ε, εγκατασταθούν. Εξαιρετική λοιπόν η πρωτοβουλία που μας προτείνεται. Thank you, Madam. Ευχαριστώ κυρία Μωρά Σαρτιέ. Ευχαριστώ πρόεδρα. Ευχαριστώ και την ε, Γκίλμετ Ντεζάν που μας παρουσίασε το Chatterbox είναι πολύ ενδιαφέρον. Εμεί στην Επιτροπή Επασχόλησης ε, συντάξαμε μία έκθεση για το θέμα ακριβώ τη επαγγελματική ένταξη των προσφύγων και υπάρχει λοιπόν συνεχώς η διαπίστωση ε, ότι θα πρέπει να δώσουμε μία όθηση ε, να επιταχύνουμε. Όπως είπε και ο συνάδελφος, όντως υπάρχει το πρόβλημα της γλώσσας, υπάρχει το πρόβλημα της αναγνώρισης των πτυχίων. Και αυτά τα δύο θέματα ε, θα πρέπει, ε, αν είχε λυθεί θα το ξέραμε, αλλά θα πρέπει να δώσουμε μία όθηση για να επιληθούν αυτά τα δύο προβλήματα και ιδίως για το θέμα της γλώσσας. Έχουμε δύο επίπεδα εκμάθησης της γλώσσας. Έχουμε μάθηση της ε, τρέχουσας γλώσσας, αυτό είναι μέρος της κοινωνικής ένταξης και την εκμάθηση της εξειδικευμένης γλώσσας για την επαγγελματική ένταξη ήδη μιλάμε για δύο είδη στόχων διαφορετικών ε, που ουσιαστικά ε, συντρέχουν προς τον ίδιο στόχο, την ένταξη, όμως θέτουν διαφορετικά προβλήματα. Το τρίτο πρόβλημα που θα πρέπει να λύσουμε όσον αφορά τη γλώσσα ε, όταν ε, πάμε στα κέντρα υποδείξης προσφύγων το βλέπουμε πολύ συχνά είναι η πολλαπλότητα των γλωσσών και θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στο ζήτημα αυτό. Αν ε, δεν υπήρχε παρά μόνο μία γλώσσα, δεν υπάρχει μία γλώσσα που μιλούν οι πρόσφυγες, προέρχονται από πάρα πολλά μέρη οι πρόσφυγες και θα πρέπει να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε πολλές γλωσσικές πρακτικές. Αυτό είναι λοιπόν ένα άλλο ζήτημα, ένα διαφορετικό θέμα με την πολυπλοκότητα που ε, ε, ενέχεται στο ότι πολλά από αυτά τα κέντρα υποδοχής προσφύγων δεν είναι και σε μεγάλες πόλεις και εγώ ξέρω πολλές ε, μεσαίες ή μικρές πόλεις όπου η ελεγγύη, η υποδοχή και η κοινωνική ένταξη μπορεί να είναι πιο εύκολες όμως η γλωσσική απάντηση είναι λιγότερο εύκολη. Έχετε σκεφτεί αυτό το πρόβλημα, έχετε κάποια στοιχεία ε, για το πώς θα μπορούσαμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό που συναντάμε επιτόπου σε ό,τι αφορά την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Αυτό που μου αρέσει πολύ στο δικό σας ε, project και που υπογραμμίζετε είναι ακριβώς ότι αφενός η γλώσσα και αφετέρου η αναγνώριση των τυχείων και η, και η επαγγελματική ένταξη θα πρέπει να επιτρέψουν ε, να έχουμε κοινωνική ανάμειξη και ε, τελικά να δούμε ότι οι πρόσφυγες κάνουν καλό στις ευρωπαϊκές μας ε, κοινωνίες γιατί δυστυχώς βλέπουμε ε, αμφισβήτηση ε, αυτού του φαινομένου της ε, κοινωνικής ανάμειξης. Εγώ θα ήθελα να μπορέσουμε να στοχεύσουμε σε αυτά τα θέματα και να τα τονίσουμε γιατί αυτό κάνει καλό και στην κοινωνία μας. Είστε έτοιμοι να απαντήσετε τις ερωτήσεις αυτές. Παρακαλώ. Να απαντήσω στα γαλλικά, μπορώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το feedback και τις ε, απαντήσεις σας. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας είπατε. Σε ό,τι αφορά την αντιστοιχεία των διπλωμάτων, των πτυχίων, ε, όταν είχα προτείνει την ιδέα αυτή, είχα γνωρίσει μια κοπέλα από την Νορβηγία που συμμετείχε σε αυτή την πρωτοβουλία. Είχε ξεκινήσει λοιπόν στην Νορβηγία για άτομα τα οποία δεν έχουν απαραίτητα πιστοποιητικό των προσόντων τους, να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να περάσουν από αξιολόγηση ευρωπαϊκό λοιπόν διαβατήριο προσόντων για τους πρόσφυγες. Το άτομο λοιπόν το οποίο θέλει να αναγνωριστούν τα προσόντα του ε, παρακολουθείται για, διάφορες, για μερικές εβδομάδες, περνάει από μια συνέντευξη και μετά μπορεί να εργαστεί στον τομέα αυτό. Είναι μια πρωτοβουλία που λειτουργεί και ξέρω ότι είναι πολύ καινούργια αυτό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, πρώτο δεύτερο έτος πρέπει να είναι. Δεν ξέρω λοιπόν πόσο επιτυχία έχει σημειώσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά ξέρω ότι χρησιμοποιείται σε επίπεδο γλωσσών. Όντως, αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Και το θέλουν. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Το θέμα των προσόντων των προσφύγων είναι ότι μπορεί να είναι χρήσιμη η εμπειρία τους. Για παράδειγμα, ξέρω ότι στον τομέα της επιστημονικής έρευνας γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτός ο κόμβος, γιατί είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει διαφορετική εμπειρία σε κάποια άτομα, σε πρόσφυγες σε ό,τι αφορά τις γλώσσες, μπορεί να υπάρχουν πρωτοβουλίες εκμάθησης της γλώσσας της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να μπορέσουν να κινηθούν και επαγγελματικά και κοινωνικά, αλλά η μητρική τους γλώσσα και η νοοτροπία τους είναι και αυτή ένα προσόν. Διδάσκω γλώσσες και σε ανήλικους και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη που έχουν ξεπεράσει το φράγμα της γλώσσας κάποια στιγμή. Για παράδειγμα, μετακομίσαμε στη Γερμανία και υπήρχαν δωρεάν μαθήματα για την δωρεάν εκμάθηση της των γερμανικών. Προφανώς η Γερμανία είναι και μια οικονομία σε καλό επίπεδο και επιτρέπει αυτό την χορήγηση δωρεάν μαθημάτων. Αλλά μου επέστησαν την προσοχή σε αυτά τα μαθήματα ευθύ εξ αρχή μόλι κατέφτασα και έτσι ξεπεράσαμε γρήγορα το θέμα του εμποδίου της γλώσσας. Θα πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε σαν προσόν το θέμα της διαφορετικής γλώσσας και στην αγορά εργασίας και στον εργασιακό χώρο. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τον κύριο Κρίστιαν Άντερσεν από τη Δανία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ε, ιδέα των οποίων λαμβάνουμε υποχρεωτικά ε, επιχειρηματικά προγράμματα στην ε, δευτεροβάθμια. Πιστεύω ότι ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα θα μπορούσε να αποτελέσει κομμάτι του προγράμματος σπουδών στα κράτη-μέλη ε, ήδη από την εφηβική ηλικία. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα προσφέρει δυνατότητες σε νέους ε, μαθητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουν γνώσεις σε τομείς όπου το πρόγραμμα σπουδών αποτυγχάνει και να τους προετοιμάσει όχι μόνο για να γίνουν μέλη μιας επιχείρησης μετά από τις σπουδέ τους, αλλά και να ξεκινήσουν μια μόνη τους. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από τρία βήματα, την παραγωγή καλών ιδεών, την εκπαίδευση για την ανάπτυξη ε, δεδομένων και τρίτον την συμμετοχή σε ε, δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης. Πρώτον, οι καλέ ιδέες δεν είναι κάτι μονάχα που υπάρχει ε, στο μυαλό κάποιων ε, σπάνιων ειδών επιχειρηματιών. Όλοι οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν ιδέες που αξίζουν να επενδυθούν, που αξίζουν να λάβουν επενδύσεις, εάν το πρόγραμμα σπουδών τους του ενθαρρύνει. Όμως, θα πρέπει να ξέρουν πώς θα προχωρήσουν με αυτό και γι' αυτό το λόγο το δεύτερο βήμα του προγράμματος θα είναι η εκπαίδευση σχετικά με το πώς να δουλεύουν με ιδέες, πώς να ανακαλύπτουν τις συγγνωμικές ιδέες, να αντιλαμβάνονται τις ε, ιδέες, ε, να ανακαλύπτουν τη βιωσιμότητα, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες. Το πρώτο και το δεύτερο βήμα μπορούν να, να, να τα επιτύχουμε δημιουργώντας ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα ε, βασίζεται σε ιδέες και προγράμματα. Θα ε, μπορούσαμε να έχουμε ιδέα για μια κοινωνική επιχείρηση η οποία θα λειτουργεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για παράγραφα. Αυτό θα συνεχίζεται καθ' τη σχολική χρονιά ούτω ώστε οι μαθητές να επικεντρώνονται σε αυτό το επιχειρηματικό έργο. Ε, τρίτον, οι μαθητές ε, με βιώσιμες ιδέες θα λαμβάνουν υποστήριξη από τα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα για να συνεργαστούν με τοπικές επιχειρήσεις και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ξεφύγουν από τα βιβλία και να πραγματοποιήσουν τις ιδέες τους. Αυτό εν τέλει θα βοηθήσει τους μαθητές ε, να εργαστούν στα δικά τους δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα προωθήσει και τι τοπικέ επιχειρήσει, συμπεριλαμβάνοντα κάτι τέτοιο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργεια των νέων στην όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσουμε οδηγίε οι οποίε ε, θα ε, προωθούν το ε, επιχειρηματικό το επιχειρηματικό πλαίσιο στο πρόγραμμα σπουδών. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιε κατευθυντήριε αντί για αυστηρά προγράμματα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. η κυρία Τλαβαγιώ αρχικά και μετά. Ευχαριστώ πολύ, Κριστιαν. Όταν μιλούσες, η εκπαίδευση ε, στα επιχειρηματικά είναι ένα μεταπτυχιακό ε, στις ήπιες δεξιότητες. Όταν μιλάμε για ήπιες ε, δεξιότητες δεν ξέρω γιατί τις αποκαλούμε ήπιες, ενώ είναι οι πιο δύσκολες να αποκτηθούν. Έχουμε συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο σχετικά με την επιχειρηματική εκπαίδευση και δεν σημαίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουμε επιχειρηματίες. Γνωρίζουμε ότι δεν γίνεται ο καθένας να γίνει επιχειρηματίας, όμως το να έχεις τέτοιες δεξιότητες σημαίνει ότι έχεις ένα καλό πλαίσιο σκέψης ε, έχω αυτούς τους ε, συνδυασμούς ε, στο κεφάλι μου. Να σκέφτεσαι έξω από τα πλαίσια, να λύνεις ε, προβλήματα, να είσαι καινοτόμος και να είσαι έτοιμος να ε, λάβεις ρίσκα. Αυτό θα πρέπει να διδάσκουμε. και θεωρώ ότι το να είσαι επιχειρηματικός σημαίνει ότι θα το, ε, θα το δούμε και στους δασκάλους και στους πολιτικούς. Όλοι οι ευρωβουλευτές που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι οποίοι είναι, έχουν επιχειρηματικό πνεύμα, διότι ε, ανυπομονούμε να ακούσουμε τις, τις ιδέες σας, είμαστε ανοιχτοί, είμαστε διατεθειμένοι να σκεφτούμε έξω από το πλαίσιο, να ακούσουμε νέες ιδέες και πραγματικά είναι μια υπέροχη ιδέα την οποία υποστηρίζω. Μου άρεσε ιδιαίτερο όταν είπες ότι θα πρέπει ε, να συνδεθούμε με ε, τοπικούς επιχειρηματίες, διότι θα πρέπει να αποκτηθούν εμπειρίες ε, στην πραγματική ζωή για τους μαθητές. Ε, αυτό είναι υπέροχο. Και επίσης λάβει υπόψη σου ότι θα πρέπει να διδάξουμε και τους ίδιους τους δασκάλους, ε, διότι για την καλή επιχειρηματική εκπαίδευση θα χρειάζεται ένας καλός δάσκαλος, ο οποίος γνωρίζει πώς θα διδάξει το μάθημα αυτό και πώς θα προετοιμάσει τις νέες γενιές για ένα τέτοιο πλαίσιο σκέψης. Έχετε λοιπόν την απολύτη υποστήριξή μου. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε μερικές ερωτήσεις παραπάνω. Το λόγο έχει η κυρία Μάκιντάιρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ιδέες σας και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η Μαρτίνα. Νομίζω ότι στην Επιτροπή Πασχόλησης μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα των νεαρών επιχειρηματιών και της υπερχηματικότητας η οποία άμα μεταφέρεται. Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι ξεκινά κανεί ε, οπωσδήποτε τη δική του επιχείρηση, αλλά είναι μια γενικότερη νοοτροπία. Υπάρχει λοιπόν ένα γενικότερο πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο στον Εμένα Βασίλειο, αλλά και σε άλλες χώρες που επιτρέπει μια ομάδα 15χρονων, 16χρονων να ξεκινήσουν μια δική τους εταιρεία. Αναφερθήκατε κι εσείς σε μια εταιρεία αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι και μια κερδοσκοπική επιχείρηση. Δεν χρειάζεται να είναι κοινωνική, κοινωνικού τύπου επιχείρηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το πρόγραμμα νεαρών επιχειρηματιών ε, σημαίνει την ε, εκλογή και ενός ε, συμβουλίου διαχειριστικού, ενός μάνατζερ και υπάρχει ανταγωνισμός υποβάλλουν τους οικονομικούς του λογαριασμού μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και οι επιχειρηματίε τη περιοχή έρχονται στη συνέχεια να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν τις πρωτοβουλίες αυτές. Πραγματικά λειτουργεί το θέμα λοιπόν αυτό και πραγματικά συμφωνώ με τη Μαρτίνα ότι θα πρέπει να διδάσκουμε και τους εκπαιδευτές γιατί συχνά οι εκπαιδευτές έχουν περάσει από μια σχολή, από το πανεπιστήμιο και στη συνέχεια έχουν συνεχίσει ως δάσκαλοι, ως ε, εκπαιδευτές στο ίδιο περιβάλλον. Αλλά κάπως θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε ως εκπαιδευτές άτομα τα οποία έχουν δουλέψει στον επιχειρηματικό κλάδο, έχουν εμπειρία, έχουν συνηθίσει να δουλεύουν με προϋπολογισμούς, ξέρω ποιοι είναι οι κίνδυνοι, οι δυσκολίες. Γιατί νομίζω ότι αν θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε το επάγγελμα των ε, εκπαιδευτών με πραγματική εμπειρία από τον χώρο εργασίας, αυτό θα βοηθούσε και το δικό σας πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Τέτσεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και ακούσαμε διάφορα σχόλια τα οποία θεωρώ θα αποβούν πολύ ωφέλιμα για τους ε, νέους που προσανατολίζονται επαγγελματικά. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι στη Γερμανία και εμείς ε, έχουμε παρόμοια εμπειρία σε ό,τι αφορά τις μαθητείες νέων, οι οποίοι πηγαίνουν σε μια εταιρεία και βλέπουν πώς ε, κινείται η ζωή στην επιχείρηση. και έτσι προσεγγίζουν την εκπαίδευση που ενδεχομένω να ήθελαν για την επαγγελματική του ζωή. Αυτό λοιπόν ε, είναι μια ευκαιρία που θα έπρεπε να τη χρησιμοποιούν όλοι οι νέοι για να αξιοποιούν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητε που έχουν προκειμένου να έχουν μια σωστή κατάρτιση. Σε τελική ανάλυση αυτό ωφελεί όμως και τις επιχειρήσεις προκειμένου να μπορούν να γνωρίζουν ε, εγκαίρως Νέου οι οποίοι από επαγγελματική άποψη και από άποψη κατάρτιση έχουν τα προσθέτα που χρειάζονται. Η κυρία Μωράν Σορτιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω είπε και η συναδέλφο Μαρτίνα Τσαμπάλαβαρ και η κυρία Μακιντάιρ, και εγώ πιστεύω ότι είναι εξαιρετικό το πρόγραμμα το οποίο συζητάμε. Αν το εξετάσουμε προσεκτικά, αποτελεί τον πραγματικό σύνδεσμο μεταξύ του κλάδου της εκπαίδευσης και του επιχειρηματικού κλάδου. Αυτό γίνεται ή με τρόπο κατακαιρματισμένο, το είπατε αγαπητέ συνάδελφε, σε ό,τι αφορά τη μαθητεία. Πρόκειται για μαθητευόμενους, εκπαιδευόμενες. Δεν είναι όλοι οι νέοι, όλοι οι μαθητές. Είτε γίνεται λοιπόν αυτό με κατακαιρματισμένο τρόπο, είτε γίνεται σε μια καθυστερήσει. Αυτό που είναι θετικό λοιπόν με το πρόγραμμά σας είναι ότι αυτή η η εξοικείωση με τις επιχειρήσεις γίνεται σταδιακά και όπως πρέπει μετά τη φάση της εκπαίδευσης με φυσικό, ομαλό τρόπο. Το δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι οι εκπαιδευτές κατά κάποιο τρόπο και αυτοί θα, θα υποχρεωθούν να περάσουν από τη δικασία αυτή, γιατί θα το ζητήσει η επιχείρηση. Είτε, είναι για, είτε πρόκειται για αναστάζ εκπαίδευση, αλλά αυτό νομίζω ότι θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την εξοικείωση με τον επιχειρηματικό κόσμο. Τι ακριβώς είναι δηλαδή ο επιχειρηματικό κόσμος, πώ αναλαμβάνονται κίνδυνοι, πώ διαχειρίζονται τα ρίσκα, πώς καταρτίζεται ένα προπολογισμό και το καθεξής. Όλα αυτά είναι προσόντα τα οποία προφανώ και μεταφέρονται. Και στο σημείο αυτό συναντάμε το πρόγραμμα το οποίο μόλις μας περιέγραψε ο Αχτούχ. Τα δύο αυτά τα προγράμματα λοιπόν είναι αλληλοσυμπληρωνόμενα. Άρα, η επιχείρηση λέτε ότι θα πρέπει να είναι μία δυτή τέτοια υποδοχή όπου μπορεί κανείς να λαμβάνει τη σωστή εκπαίδευση και αυτό που προτείνετε εσείς είναι να υπάρχουν αυτά τα προσόντα τα οποία μεταφέρονται, το οποίο και θα επιτρέψει να προωθηθεί η κινητικότητα σε επαγγελματικό επίπεδο από τη μία θέση στην άλλη. Αυτό άλλωστε είναι και ο καλύτερος εξοπλισμός, αν θέλετε, του ατόμου, του επαγγελματία απέναντι στην ανεργία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι δύο από τα τρία αυτά προγράμματα που απευθύνονται και στο γενικό πληθυσμό, χωρίς να υποβιβάζω το πρόγραμμα σας για τους πρόσφυγες, έχουν ένα πραγματικά έντονο σύνδεσμο μεταξύ τους. Και ασφαλώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και να βρούμε με τέτοια σύνδεση και με το πρόγραμμα για τους πρόσφυγες. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο θα υπερνικήσει τις, ε, τα εμπόδια που έχουμε αυτή τη στιγμή, όπου τα πράγματα είναι κατακαιρματισμένα και η επαγγελματική εμπειρία έρχεται πολύ καθυστερημένη. Γι' αυτό άλλωστε εκκινήσαμε και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, για να δώσουμε απαντήσεις σε τέτοια ζητήματα. Αλλά εσείς με το πρόγραμμά σας ε, δίνετε τις απαντήσεις και τις λύσεις από την ρίζα του προβλήματος. Γι' αυτό λοιπόν και σας συγχαίρω και σας ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Μαρτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω κι εγώ. Δηλαδή να μάθουν οι νέοι από το σχολείο ήδη τον επιχειρηματικό κόσμο και γιατί όχι μπορεί να θέλουν και να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Πολύ ωραία λέγω. Νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο τους νέους, αλλά όλα τα κοινωνικά τα στρώματα. Εδώ ψηφίζουμε νόμου που έχουν αντίκτυπο στην επιχείρηση και πολλοί δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στι επιχειρήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, παραδείγματο χάρη, θα σα ε, αναφέρω τέσσερα παραδείγματα για την ε, ε, έχουμε έναν επίτροπο για την ενέργεια, τη βιομηχανία και τα λοιπά Άλλον για τον ανταγωνισμό, άλλον ε, για την απασχόληση. Ε, δηλαδή έχουμε τέσσερις επιτρόπους για τέσσερα οριζόντια ζητήματα που αφορούν το επιχειρηματικό κόσμο. Και όταν μιλάτε για έναν επίτροπο για ένα θέμα θα σου πει «Α, δεν είναι δίκες προποδιότητες αυτό και αυτό πρέπει να το πλουστεύσουμε». Δηλαδή όταν θέλουμε να ψηφίσουμε νόμους και θέλουμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο όραμα, τότε ε, πρέπει να ξέρουμε ότι και μια επιχείρηση δεν είναι κατακαιρματισμένη. Μια τέτοια επιχείρηση ε, που θα έχει στεγανά, ε, τότε θα οδηγηθεί στην αποτυχία. Όμως ε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν όλα αυτά και ίσως θα πρέπει να έχουμε ένα και μόνο επίτροπο για αυτούς τους τέσσερις μεγάλους φακέλους που αφορούν γενικά τον επιχειρηματικό κόσμο. Πολύ ωραία είναι η ιδέα. Και εγώ έχω κάνει μια σχετική κατάρτιση και ακόμη και πιο έρχομαι από τον επιχειρηματικό κόσμο. Υπήρχαν ε, όμως ε, πολλοί άλλοι εκλεγμένοι αιρετοί που ανακάλυπταν μαζί μου τον επιχειρηματικό κόσμο. Έτσι λοιπόν εγώ θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να απευθυνθούμε στην κοινωνία. Yeah, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και σας ευχαριστώ που Αναγνωρίσατε το νόημα της ιδέας σε ό,τι φορά τώρα τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών, γιατί πολύ αναφερθήκατε σε αυτό, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Νομίζω μία προσέγγιση θα ήταν όχι μόνο να πάρουμε τους μαθητές από την αίθουσα και να τους βάλουμε στις επιχειρήσεις όπως προτείνεται με τις μαθητείες, αλλά να φέρουμε και τις επιχειρήσεις μέσα στην αίθουσα συμπεριλαμβάνοντας ε, τοπικούς επιχειρηματίες ε, στην αίθουσα έτσι ώστε να μπορούν απευθείας να έχουν λόγο στην εκπαίδευση. Και συμφωνώ με τον κύριο Μαρτά. Είναι σημαντικό να ανοίξουμε τα μάτια μας ε, σε αυτή την προοπτική και μου αρέσει πραγματικά ο σύνδεσμος μεταξύ της ιδέας του Άρθουρ και της δικής μου Βλέπω ότι υπάρχουν στενοί σύνδεσμοι. Ευχαριστώ. Ε, the Ίσως η Κομισιόν ε, θέλει να αντιδράσει, να συνοψίσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είχα ε, κατά νου το πρώτο και το τρίτο project που πραγματικά συνδυάζονται πολύ καλά. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία του Junior Achievement που ουσιαστικά ε, αφορά στο να συστήνονται φοιτητικέ εταιρείε σε διάφορε χώρε και αναφέρθηκε η κυρία Μακιτάιρ σε αυτό το θέμα. Ε, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι εμπνέονται να συστήσουν μια εταιρεία ε, και να τη δικήσουν και αυτό είναι μια καλή αρχή. Αλλά να έχουμε μια οριζόντια κατάρτιση για την επιχειρηματικότητα, αυτό δεν υπάρχει ακόμα γιατί σήμερα συμμετέχουν πολύ λίγοι μαθητές 15-16 χρονών. Η κατάρτιση για την επιχειρηματικότητα είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε όσο δυνατόν περισσότερο κάτι τέτοιο Δηλαδή όχι μόνο ε, σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και στη γενική εκπαίδευση, γιατί οι άνθρωποι που έχουν ιδέες μπορούν αργότερα να λάβουν και κάποια οικονομική στήριξη που θα παρέχεται από διάφορα ευρωπαϊκά μέσα, παραδείγματος χάρη το μέσο ε, για τα ε, μακροοικονομικά που υπάρχει σε πολλά κρατημέλη, υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο μέλλον. Και επίσης μεταξύ των προσφύγων ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μαθητεία γιατί υπάρχουν κάποια πιλωτικά προγράμματα που προετοιμάζονται και εφαρμόζονται υπό το πρόγραμμα COSME για την υποστήριξη στις ΜΜΕ και το πρόγραμμα καινοτομία να βοηθήσουν τους, που βοηθούν τους πρόσφυγες ε, για να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση. Ε, γιατί είναι δύσκολη η πρόσβασή του στη χρηματοδότηση, ακόμη και αν έχουν την καλύτερη ιδέα. Έτσι, λοιπόν, αυτά τα μέσα υποστηρίζουν του πρόσφυγε να ξεκινήσουν τι επιχειρήσει του και να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά του προσόντα και να αντεχθούν ευκολότερα στην κοινωνία. Μου αρέσουν, όλα τα project. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιο είναι καλύτερο, κάποιο χειρότερο. Χαίρομαι πολύ που να μα παρουσιάζουν αυτέ τι ιδέε και πραγματικά αισθάνομαι καλά που κάποιο από το δικό μα σκεπτικό επίση οδεύει προ αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν μόνο το πρώτο μέρος. Τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Άρθουρ. Μας παρουσιάσει κάποιες ιδέες, ίσως και κριτικές, για το Erasmus Change some Θέλεις να γίνουν κάποιες αλλαγές. Παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η δεύτερη πρόταση που παρουσιάζω ε, η έκκληση να δράξουμε την ευκαιρία που προσφέρει το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, ο σχεδιασμένη διπλασιασμό χρηματοδότηση για το Erasmus Plus ε, θα πρέπει να χρησιμεύσει για να προωθήσουμε την κινητικότητα εκμάθηση ένταξη, αυξάνοντα την υποστήριξη για την διεθνική εκπαίδευση και κατάρτιση παρά τις, ε, τις προσπάθειες ε, που γίνονται μέσω του Erasmus Pro και του Mobility της χάρτες για την κινητικότητα, η, κινητικότητα παραμένει περιθωριακή. Μόνο το 17% των ευκαιριών Erasmus ε, αφορούν τους φοιτητές επαγγελματική εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μου. Έχουμε μόνο 8 κατόχους της χάρτας που παρέχουν ευκαιρίες για τους φοιτητές ταυτόχρονα. Ε, είδαμε ότι ε, Λιγότερο από το ίμιση των 7.100 αιτήσεων για επαγγελματική και κατάρτιση πήραν χρηματοδότηση, ε, ενώ το 97% στην άνωτερη εκπαίδευση έλαβαν. Αυτό είναι απογοητευτικό όταν αναφερόμαστε στην παράδοση ε, της ε, Ευρώπης για τη μαθητεία στο εξωτερικό. Γιατί όχι λοιπόν σήμερα θα πρέπει να έχουμε περισσότερες προσπάθειες να διευρύνουμε τους χρηματοοικονομικούς πόρους στο Erasmus+, ενώ θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης, διασφάλισης ποιότητα και διαφάνεια. Πολωνίας μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστοτικών Ομάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ε, την ε, Ευρωπαϊκή Διασφάλιση Ποιότητας και το πλαίσιο ε, ευρωπαϊκών προσόντων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια ισχυρή δέσμευση οικονομική για να δείξει πολιτική βούληση, να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για κινητικότητα ΒΕΤ. Τα νέα μέσα από το Erasmus Plus θα πρέπει να αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας για τις αιτήσει ΒΕΤ για να υποστηρίξουμε του ε, μαθητέ ε, κυρίω ε, που προέρχονται από μειονεκτικέ ομάδε. για να αυξήσουμε το ποσοστό επιτυχία και οι εταιρείε και όσοι υπάροχοι επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να ενταχθούν στο οικοσύστημα του Erasmus Plus αυξάνοντας τον αριθμό των υπογραφώντων στην χάρτα κινητικότητας. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει και την καταλληλότητα των αιτήσεων η ανοιχτή διαβούλευση για το Erasmus Plus έχει δείξει ότι ένα συγκεκριμένο εμπόδιο στην κινητικότητα προκύπτει από το κόστος ε, που έχουν οι εργοδότες για να προωθήσουμε την χάρτα κινητικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων ε, θα πρέπει η χρηματοδότηση να επιδοτεί την απασχόληση για τους ε, μετακινούμενους μαθητευόμενους. Οι νέοι ε, είναι φιλοευρωπαίοι χάρη στις ευκαιρίες που τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους βοηθήσουμε όλους να υποφεληθούν άμεσα από μια ευρωπαϊκή κοινωνική διάσταση. Αυτή είναι η ευκαιρία που έχετε τώρα. Να την αδράξετε. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λαπετσόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι ακριβώς ε, είναι σαν να διαβάζετε το μυαλό μου, τις σημειώσεις μου. Ήμουνα από του ευρωβουλευτέ που πριν από τρία χρόνια ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για ένα νέο εράσμο για σχολεία επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και πραγματικά βίωσα αυτά ε, τα οποία ε, είπατε. Αρχικά λοιπόν στην Ευρώπη έχουμε διαφορετικά συστήματα επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οπότε το να έχουμε μια κοινή χάρτα και να επιτρέπουμε την, ε, την απόκτηση εμπειρίας μέσω τη κινητικότητα. στα διάφορα διάφορα κράτη-μέλη θα ήταν κάτι υπέροχο. Μπορώ να σας πω από εμπειρία ότι στη χώρα μου, την Τσεχία, ε, είμαστε πολύ συνδεδεμένοι με την ε, Γερμανία λόγω της οικονομίας, των εξαγωγών, εμπόριο, επενδύσεις. Ε, όμως το διαδικό σύστημα της Γερμανίας δεν ταιριάζει με το τσεχικό εκπαιδευτικό σύστημα, οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε τη δική σας χώρα, την Αυστρία, διότι είναι ένας διαφορετικός τρόπος εφαρμογής του διαδικού συστήματος, του διοικού συστήματος, Οπότε πιστεύω ότι είναι το ιδανικό. Έχω τρία σημεία τα οποία πιστεύω ότι είναι δύσκολα στην ε, περαιτέρω ανάπτυξη του, ε, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ε, στο πλαίσιο Εράσμου. Το πρώτο πρόβλημα είναι η κοινή αναγνώριση, πάνω στο οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεύτερον, η γλώσσα η ε, μάθηση, ε, εκμάθηση ξένων γλωσσών σε τέτοια σχολεία δεν είναι κάτι τόσο σύνηθες όσο είναι στα πανεπιστήμια. Οπότε ίσως αυτό να είναι ένα πρόβλημα, οπότε θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερα γλωσσικά μαθήματα. Και τρίτον, ε, πρακτικό ότι μερικές φορές οι μαθητές δεν βλέπουν ε, τη δυνατότητα, δεν βλέπουν ε, κάποιον ε, που να είναι διαχειριστής τέτοιου προγράμματος σε επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που να είναι υπεύθυνο να διαχειριστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Φανταστείτε, όταν έγινε το, το κάλεσμα για το Εράσμους ε, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εγώ έστειλα ε, σε 750 τέτοια σχολεία στην Τσεχία επιστολές για να τους δώσω αυτή την πληροφόρηση. Υπάρχει νέα κλίση, νέο ε, περίοδος αιτήσεων και το αποτελέσμα όλα σχεδόν ρωτούσαν από το δικό μου γραφείο να τους κάνει τη διαβούλευση για την αίτηση διότι δεν, ήξε, δεν είχαν κάποιον project manager στα σχολεία τους. Οπότε θα πρέπει να επιληθεί και αυτό το θέμα. Θα πρέπει να γίνει πιο εύκολο για τα σχολεία να μπορούν να κάνουν αίτηση και να εργαστούν σε ε, διεθνή προγράμματα. Παρ' όλα αυτά όμως πολύ καλή ιδέα. Άρτουρ, πιστεύω ότι πρέπει να έρθει να δουλέψει για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο στον κύριο Ντέτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ε, χαιρετήσω εκ μέρους της συναδέλφου Άγνες Γιονκέριους η οποία σήμερα έπρεπε να είναι ε, στη συνάντηση των σχεδιών ε, για το ζήτημα του προϋπολογισμού όχι μόνο να διπλασιαστεί αλλά να τριπλασιαστεί ο προϋπολογισμός για αυτό το θέμα και αυτή είναι η θέση των δημοκρατών. Νομίζω ότι είναι εκ των όνων κάνευ ότι στην επαγγελματική εκπαίδευση, να επενδύσουμε ε, περισσότερο και να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς να βγουν από τη χώρα τους ε. και μιλήσατε επίσης ε, για τα χρόνια μαθητείας ε, τα οποία υπάρχουν ε, στις γερμανόφωνες ε, χώρες και από ό,τι ακούω φτάσανε μέχρι και τη Γαλλία. Πιστεύω λοιπόν ότι το ερώτημα των ταξιδιών σε συνάρτηση με τη μαθητεία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε θετικά εάν το υποστηρίξουμε αυτό και το ενσωματώσουμε στην επαγγελματική κατάρτιση των ανθρώπων αρχής εξ αρχής και ξεκαθαρίσουμε ότι κομμάτια της επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να γίνουν και σε γειτονικέ χώρες και έτσι δίνεται η δυνατότητα να συνεχιστεί και να συμπληρωθεί η εκπαίδευση κάποιου σε μια γειτονική χώρα. Θα ήθελα επίσης ε, να δω αν ελέγχατε κατά πόσο, κατά πόσο οι επιχειρηματίες, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να, να συνεισφέρουν σε όλο αυτό, ούτως ώστε ε, οι νέοι αρχής εξ αρχής να έχουν την δυνατότητα ε, και μέσω ε, συγκεκριμένων προγραμμάτων ε, να προσθέτουν στην εκπαίδευσή τους και γλωσσικά μαθήματα και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν αυτό στην Ευρώπη, το πώς ε, θα μπορέσει να υπάρχει μια σύγκληση της αναγνώρισης των διαφόρων σημείων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να δούμε τις ε, θετικές δυνατότητες που υπάρχουν για τους ε, νέους όταν στο πλαίσιο της εκπαίδευσή τους ε, πηγαίνουν και σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα φέτος είδα το, στις Βρυξέλλες το πρόγραμμα όπου υπήρχε μια ανταλλαγή μεταξύ Ισπανίας, Ιταλίας, και Γερμανίας ε, και θα πρέπει να δούμε λοιπόν το πώς ε, και σε άλλες χώρες θα δοθούν οι δυνατότητες σε νέους ε, για ένα μήνα έστω κομμάτι της εκπαίδευσής τους να την κάνουν σε άλλη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να εξισορροπηθεί, να γεννήσει με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πολύ καλή δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτό και στις σπουδές μου καλύπτουμε στο Πανεπιστήμιο τα συγκεκριμένα θέματα, το ζήτημα της κοινή αναγνώρισης, και, τις, και τα διάφορα συστήματα που υπάρχουν, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται και δείχνουν το πόσο μειονεκτό τα, ε, τα σχολεία επαγγελματική εκπαίδευση ε, στην απόκτηση χρηματοδότηση και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Όπως επίσης το γεγονό ότι αυτά τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν στην χάρτα κινητικότητα έχουν ένα ε, ποσοστό επιτυχίας 97 με 98% ε, στις αιτήσει τους, το οποίο σημαίνει ότι είναι απλά ένα ζήτημα χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα όμως οι αιτήσει ε, δεν είναι επαρκείς. Δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση για τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν στο οικοσύστημα του Erasmus Plus και θα πρέπει λοιπόν να ενσωματωθούν σε αυτό το σύστημα. Όταν μιλάμε λοιπόν για τους λόγους που όλο αυτό έχει σημασία, Υπάρχει φυσικά το θέμα της ε, αυτοβελτίωσης, η μάθηση, εκμάθηση γλωσσών, οι βασικές δεξιότητες, οι ποιες ικανότητες, ε, όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα, όμως υπάρχει και η λειτουργική αξία από άποψη πολιτικής, ε, το οποίο πιστεύω ότι δεν αναφέρεται συχνά και αφορά την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου από νέους ένας στους δέκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, σπουδάζουν, σταματούν ε, το σχολείο. Πολλοί μεταξύ 19 και 16 και 19 ετών ε, συμμετέχουν, είναι μέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οπότε το πρόγραμμα INVET έχει μια έκθεση η οποία λέει για ποιο λόγο οι νέοι εγκαταλείπουν ε, τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ένας λόγος είναι ότι υπάρχει έλλειψη επαγγελματικής προοπτικής και, προσωπική, και προσωπικό κίνητρο για να ε, συνεχίσουν περαιτέρω στην επαγγελματική εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν η προοπτική του να βγουν στο εξωτερικό, να ε, βελτιωθούν ακόμα πιο πολύ, μπορεί να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα τα οποία ίσως να μην σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Η κυρία Μωρασέτια. Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά είπε ο Άρθουρ κάτι πολύ σημαντικό. Ότι πολύ συχνά το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Erasmus Plus ε, ε, αφορά ανθρώπους που είναι ήδη σε κατάρτιση. Εγώ προωθώ την γεωγραφική κινητικότητα για νέους που έχουν βγει από τα εκπαιδευτικά συστήματα χωρίς ε, κάποιο τίτλο. Γιατί το σημαντικό για αυτή τη γεωγραφική κινητικότητα είναι να μπορεί κάποιος ε, να είναι περήφανος για την ενοικοδόμηση του εαυτού του και αυτός είναι ο πυλώνας βάσει του οποίου μπορεί να οικοδομήσει κάποιος και στο πλαίσιο των νέων και για τους νέους που έχουν βγει χωρίς ε, κάποιο τίτλο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή να πάρουμε τους νέους ε, που δεν έχουν ε, προσόντα, που έχουν χάσει την αυτοπεποίθησή τους, έχουν χάσει την εικόνα του εαυτού τους και να τους εμπλέξουμε στην κινητικότητα σε οποιοδήποτε κλάδο και ακόμη και αν δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας όπου θα πάνε, Παραδείγματο χάρη από τη Γαλλία μπορούν να πάνε άνθρωποι στην Ελλάδα, στη Λιθουανία, στην Ισπανία. Ε, έχω στείλει εγώ ανθρώπου από το κέντρο τη Γαλλία εκεί. Πήγαν και επέστρεψαν και ήταν περήφανοι και είχαν ε, όρεξη και στο τέλος τη κατάρτισής τους είχαν και κάποιες ιδέες για συγκεκριμένα προγράμματα, για συγκεκριμένα project. Έτσι λοιπόν αυτή η οικοδόμηση είναι πολύ σημαντική. Και θα πρέπει να ξέρουμε να στηριχτούμε σε αυτό. Το δεύτερο σημείο, είπατε, δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφοι. Είναι σίγουρο ότι και στους νέους και τους νέους, όπως και τους ενήλικες, τους φοβίζει η κινητικότητα και για να βρούμε ένα παράγοντα που να άρει το φόβο αυτό νομίζω ότι πρέπει να προωθήσουμε το γεγονός ότι όλοι οι λέει που έχουν ε, πάει σε προγράμματα ή έχουν συμμετέχει σε προγράμματα επαγγελματική, ε, συγγνώμη, γεωγραφικής κινητικότητας, διορθώνω μιλήτρια, μπήκαν ε, στην αγορά εργασίας πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας επιταχυντής εδώ και πρόκειται για νέους που αντιστέκονται καλύτερα στην ανεργία γιατί στη γεωγραφική κινητικότητα ουσιαστικά αντιστοιχεί και επαγγελματική κινητικότητα. Δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πολύ θετικά επιχειρήματα έτσι ώστε περισσότεροι νέοι να θέλουν να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα κινητικότητας. Είναι ένα συν της Ευρώπης. Προγράμματα όπως το Erasmus Plus, ε, σε όλους μπορείτε να μιλήσετε, σε οποιοδήποτε ε, όλοι τα γνωρίζουν, όλοι έχουν ακούσει να μιλάνε για το πρόγραμμα αυτό. Και θα πρέπει όχι μόνο να αυξήσουμε τον προπολογισμό όπως έχουμε κάνει, και για μένα είναι μια γραμμή του προπολογισμού που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί εδώ έχουμε βιώσιμα αυτά αποτελέσματα επί της απασχόλησης και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτός ο πολύ θετικός για να έχουμε περισσότερους συμμετέχοντες, περισσότερους υποψήφιους στο πρόγραμμα αυτό. Thank you. Um... Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, Γκουγιμέτ uh, Tijan. Ευχαριστώ πολύ. Η δεύτερη μου ιδέα είναι η δημιουργία ε, μιας, ε, ένα, ενός ευρωπαϊκού ε, προγράμματος επιχειρηματικών φυτορίων για μετανάστες που θα τους προσφέρει καθοδήγηση για τη δημιουργία επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν βοήθεια στη συνέτησή τους για λήψη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και θα λαμβάνουν διοικητική και νομική υποστήριξη. Αυτά θα βοηθήσουν να ενσωματωθούν οι μετανάστες, οι πρόσφυγες στην κοινωνία κοινωνία, όχι μονάχα μέσω της απασχολησιμότητας, αλλά και με τη δημιουργία βιώσιμων μηχανισμών απασχόλησης. Ταυτόχρονα θα δημιουργήσει ποικιλία στην ε, ευρωπαϊκή επιχειρηματική αγορά. ενώ από τα πιο σημαντικά ζητήματα για την κοινωνία μας σήμερα είναι οι νησότητες, στις οικονομικές δυνατότητες. Η επιχειρηματικότητα είναι ένας αποτελεσματικό μηχανισμός ε, για την κινητικότητα και ιδιαίτερος ε, για πληθυσμούς οι οποίοι φέρουν στίγμα. Δυστυχώ όμως για ανθρώπους με προσφυγικό υπόβαθρο υπάρχει ένα μεγάλο επιχειρηματικό χάσμα και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δεν έχουν πρόσβαση ε, σε ε, δίκτυα επιχειρηματικότητας ε, και επενδύσεων, ε, δεν έχουν πρόσβαση σε διοικητικές και νομικές διαδικασίες και βοήθεια, το οποίο αποτελεί ένα εμπόδιο, δεν γνωρίζουν την κοινωνία, δεν γνωρίζουν τις διοικητικές διαδικασίες με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να κάνουν λάθη που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Και επίσης έχουν ε, ελπί πρόσβαση σε δυνατότητες ανταλλαγή δεξιοτήτων. Τα φυτώρια αυτά θα αυξήσουν την δυνατότητα για την επιτυχία των επιχειρήσεων, έχουν ένα ποσοστό ε, βιωσιμότητα 87%, ε, ενώ οι επιχειρήσεις που δεν έχουν βοήθεια έχουν ποσοστό επιτυχίας μόνο 44%. Τα προγράμματα αυτά υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Η Πατριαρμοστία του ΟΗΕ έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα στο Εκουαδόρ, στον Ισημερινό το 2011 ε, το οποίο έδωσε την δυνατότητα σε πρόσφυγες να δημιουργήσουν επιχειρήσεις ακόμα και σε ε, περιοχές που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες. Ε, και βλέπουμε ότι ακόμα και στην Νορβηγία αυτή τη στιγμή η Startup Refugees έχει υποστηρίξει 60 επιχειρήσεις τις οποίες διοικούν οι πρόσφυγες και έχει προσφέρει 4.000 μαθήματα τα οποία ε, τους έδωσαν την δυνατότητα ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Ε, επίσης, αυξάνουν τις δυνατότητες αποσχολησιμότητας για άλλους ε, πρόσφυγες και αποτελούν έναν επιτυχημένο μηχανισμό για την καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον αυτών των πληθυσμών. Ε, βίωσα αυτή την επιτυχία με την ε, ε, Μουσάλ Χεντεγιάτ, η οποία είναι η ίδια πρόσφυγας και με την οποία συνειδρήσαμε πριν από δύο χρόνια το Chatterbox για να βοηθήσει τους πρόσφυγες ιδρύθηκε από επενδυτές που προσπαθούν να κάνουν επιρροή και γεφύρωσε τα χάσματα τα οποία ανέφερα προηγουμένως, τα οποία πολλές φορές είναι αόρατα. Ε, έτσι έδειξε τη δυνατότητά του, κέρδισε εμπιστοσύνη και έδειξε το πώς μπορεί να ενώσει τις κοινότητες με ε, επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή έχει χρηματοδοτική υποστήριξη από την Silicon Valley και έτσι λοιπόν μπόρεσε να αναπτυχθεί ως ε, επιχείρηση και να βοηθήσει την κοινωνία. Ένα τέτοιο φυτόριο θα προσφέρει δυνατότητα πρόσβασης ε, σε χρηματοδότησης ε, καθώς επίσης και δυνατότητες όσον αφορά την, ε, τις δυνατότητες μαθητείες, ειδίκευσης, θα γκρεμίσει τα, όρ, τα, τα φράγματα, θα δώσει τη δυνατότητα τους, τους πρόσφυγες να γίνουν οικονομικοί παράγοντες της νέες κοινωνίες και θα δώσει την δυνατότητα στην δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καινοτόμου επιχειρηματικού χώρου. Πιστεύω λοιπόν ότι τέτοιες επιχειρήσεις ε, εποφελούν, βοηθούν ε, στην ε, σχέση μεταξύ των προσφύγων και των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Detchen. Ο κύριος Είμαι ενθουσιασμένος από τις ιδέες που άκουσα από την κυρία Ντεζάν, διότι Πίσω από αυτό κρύβεται ένα πολύ μεγάλο δυναμικό το οποίο πρέπει άμεσα να χρησιμοποιήσουμε στην Ευρώπη να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους ε, ώστε να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι χωρίς να χρειάζονται βοήθεια, με τις ικανότητες τις οποίες φέρνουν από τις πατρίδες τους, τις οποίες έπρεπε να εγκαταλείψουν, έχουν τώρα την δυνατότητα ε, με λίγο κεφάλαιο να δημιουργήσουν μια νεοφυή επιχείρηση. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, το Chatterbox ε, είναι κάτι ε, υπέροχο διότι μπορούμε να βοηθήσουμε με την εκμάθηση γλώσσας για παράδειγμα όπως αναφέρατε. Υπάρχουν πολλές άλλες δεξιότητες και εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε σχετικά με το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τέτοια προγράμματα ούτως ώστε να αποτελέσουν πρότυπα και στη συνέχεια. Το θεωρώ πραγματικά υπέροχο και ευχαριστώ πολύ για τα συγκεκριμένα κίνητρα. Thank you. Do Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε, να αντιδράσετε. Ναι, πολύ σύντομα. Σίγουρα, βεβαίως, θα ήθελα να συζητήσουμε ευρύτερα αυτό το project. Εγώ φυσικά πρέπει να κάνω πολλή έρευνα λόγω της δουλειάς μου σε αυτό. δεν ε, υπάρχουν πολλές μελέτες γιατί αλλάζουν συνεχώς τα νούμερα. Παραδείγματος χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 20% του πληθυσμού των ε, προσφύγων ε, έχουν προσόντα ενώτα της εκπαίδευσης, όμως είναι τεράστια η ενεργεία και πολλοί μπορεί να είναι και επικεφαλής σε επιχειρήσεις, επομένως χάνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες και θα ήθελα να συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το ζήτημα. Κυρία Μωρανσαρτιέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στον αντίδραση του συναδέλφου. Και εμένα μου αρέσουν πολύ οι που προτείνετε. Και επομένως ε, έχω μπει σε προβληματισμό ε, σε σχέση με το πώς θα τεθούν σε εφαρμογή για το επόμενο στάδιο δηλαδή. Ένα ζήτημα που με ανησυχεί είναι το θέμα της εδαφικότητας. Συχνά τα κέντρα προσφύγων, όπως είπα και πριν, βρίσκονται σε μικρές ή μεσαίες πόλεις. Δεν είναι απαραίτητο σε μεγάλες πόλεις. Επομένως, πώς θα συσχετίσουμε ε, τη δημιουργία αυτού του φυτορίου ε, με την γεωγραφική κατανομή των προσφύγων στη Γαλλία, στη χώρα μου. Τα κέντρα υποδοχής προσφύγων ε, είναι πάρα πολύ διάσπαρτα και τα εκολαπτήρια κυρίως υπάρχουν σε πανεπιστημιακές πόλεις όπου υπάρχει ένα τεχνολογικό δίκτυο επιχειρήσεων σε μεγαλύτερη συγκέντρωση. Έχετε σκεφτεί συστήματα ε, εξαποστάσεως ε, κατάρτισης. Δηλαδή πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αφενός έχουμε τα κέντρα προσφύγων που είναι διάσπαρτα στην επικράτεια και έχουμε από την άλλη αυτά τα κολαπτήρια που είναι σε μεγάλες πόλεις πανεπιστημιακές. Ε, και έχετε σκεφτεί ένα τέτοιο μηχανισμό. Φαντάζομαι όμως ότι εσείς δεν θέλετε να επικεντρωθείτε μόνο σε μεγάλες πόλεις. Ε, φαντάζομαι σκέφτεστε να υποφεληθούν όλοι. Έχετε σκεφτεί κάποιες τεχνικές, πώς μπορούμε λοιπόν να ε, παρακάμψουμε αυτό το γεωγραφικό πρόβλημα. Απάντηση. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να πάρουμε αυτά τα εμπόδια, αυτούς τους περιορισμούς ε, και να τα κάνουμε πλέον κτήματα, δηλαδή ε, τους χάρη όλοι οι συμμετέχοντες να συμμετέχουν σε τοπικό επίπεδο και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο. τους χάρη μπορούμε να έχουμε και κάποιους καθοδηγητές, μέντορες, ε, επενδυτές. Νομίζω ότι το κεφάλαιο μπορεί να έρθει από ε, ευρωπαϊκά κονδύλια και από τις ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά μπορούν να συμμετέχουν και επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για να συνδεθούμε τοπικά και ουσιαστικά ε, να μπορέσουμε να κάνουμε τον ε, επιχειρηματικό και κοινωνικό ιστό πιο ανθεκτικό σε όλη τη χώρα. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Κριστιαν. Ευχαριστώ πολύ. Η δεύτερη ιδέα μου είναι ε, να βοηθήσουμε τα επαγγελματικά ιδρύματα να παρέχουν επαρκείς ευκαιρίες μαθητείας σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες προκειμένου να δίνουν ε, επαγγελματικό προσανατολισμό σε νέους και να αντιμετωπίσουν ε, τα ποσοστά ενεργείας των νέων. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγήσει κονδύλια ε, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνε ε, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όταν ε, θεσπίζουν και δικούν μαθητείε. Είναι μια σημαντική απόφαση, τολμηρή απόφαση για του εργοδότε να προσλάβουν ένα νέο χωρί εμπειρία και δεν είναι όλοι οι εργοδότε τολμηροί και γιατί θα πρέπει να επιλέξουν ένα νέο χωρί καθόλου πείρα αντί πιο πεπειραμένου, ε, βελτιώνοντας ε, τις ε, ευκαιρίες κατάρτισης και μαθητείας, ναι, θα είναι πιο έμπειροι και θα μπορούν να είναι πιο ελκυστικοί για τους εργοδότες. Σε μελλοντικέ συνεντεύξεις, ο πιθανός εργοδότης θα ξέρει ότι ο υποψήφιος είναι κάποιος που έχει ήδη κάποια πείρα αυτό θα είναι πλεονέκτημα για τους νέους που προσπαθούν τώρα να βρουν δουλειά. Φαντάζομαι ότι μία περίοδος μαθητείας θα είναι έντονη και σύντομη έτσι ώστε να μπορεί να ενταχθεί σε ένα σχολικό πρόγραμμα ακόμη και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από την ηλικία των 8. Η ερώτηση που πρέπει να τίθεται είναι τι θέλεις να κάνεις, όχι τι θες να γίνεις. Θα μπορούσαν να διαρκούν οι περίοδοι αυτοί από μία σε δύο εβδομάδες ανάλογα με το πρόγραμμα και θα λάμβαναν χώρα άπαξ ετησίω. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα σχεδιάσουν ε, του μαθητείε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για κάθε μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι κάποιε μαθητείε θα διαρκούν ολόκληρη τη μέρα, ενώ άλλε θα είναι λίγε ώρε εργασία ε, και κατόπιν θα συνεχίσετε το σχολικό πρόγραμμα. Από τη σκοπιά των επιχειρήσεων ε, που συμμετέχουν σε τέτοιες συνεργασίες με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι, ε, οι δεν θα πληρώνονται, έτσι λοιπόν θα είναι πιο ελκυστικό για τις επιχειρήσεις. Έχω φίλους στη Γερμανία και στη Σουηδία που αποφάσισαν ότι αυτό που θέλουν, αυτά που θέλουν να πετύχουν στην καριέρα τους σε βάση εμπειριών ε, σε περιόδους μαθητείας. Έτσι λοιπόν η πρόταση αυτή, πέρα από το να μειώσει την ενεργεία των νέων, θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να καλύψουν οι μαθητές ε, τι τους αρέσει και ποιοι επαγγελματικοί τομείς μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για αυτούς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας ε, επιδοτήσεις ε, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θέλουν να παρέχουν στους μαθητές τους την ευκαιρία αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει το λόγο του Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ανέφερα ότι όλα τα προγράμματα που διάβασα, ακόμα και οι τίτλοι τους είναι ενδιαφέροντες. Και αυτό επιβεβαιώνει εκ νέου ότι χρειαζόμαστε πολλές εταιρικέ σχέσεις. Για όλες τις ιδέες που, παρε... παρουσιάσετε σήμερα, χρειαζόμαστε συνεργασίες. Συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των πολιτικών ηθινόντων. Επίσης, πιστεύω ότι στην ιδέα της μαθητείας για να διευρυνθεί στο βαθμό του δυνατού η έννοια της μαθητείας απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτό αποτελεί και στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων να εντοπιστούν διάφοροι παράγοντες. Καταρχάς, κατά πόσο πρόκειται για το σωστό μέρος για τους ε, νέους. Τι θέλουν να πετύχουν και να βοηθήσουμε να μάθουν τα άτομα αυτά τι σημαίνει η δουλειά ακριβώς, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ε, ε, είναι δύσκολο για τους νέους τους παίρνει κάποια χρόνια, κάποιο χρόνο να προσαρμοστούν στην ιδέα της εργασία και το πώς ακριβώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται και την ε, πειθαρχία που θα πρέπει να επιδείξουν. Είναι σημαντικό βήμα αυτό λοιπόν. Το 2013 υπογράψαμε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Μαθητείες ε, σε 26 κράτη-μέλη υπάρχουν ε, κάποιες χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν ε, δεσμευτεί να δώσουν 900.000 θέσεις για μαθητεία. Πριν από 10 μέρες ε, έγινε τρίτη εβδομάδα για την επαγγελματική κατάρτιση η οποία αναφέρθηκε ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία από πλευρά των επιχειρήσεων για τις μαθητείες και για να συμμετάσχουν στις στην χορήγηση ικανότητων προς τους νέους, χορήγηση ικανότητων και προς που θα χρειαστούν στο μέλλον της επαγγελματική τους ε, ζωής. Θα ήθελα να σχολιάσω και να πιστήσω την προσοχή σε ένα πλατικό πρόγραμμα, το Erasmus Pro, το οποίο ξεκίνησε ως πλατικό πρόγραμμα στους κόλπους του Κοινοβουλίου και πλέον καθιστεται βασικό πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Erasmus Plus ε, που και δίνει ε, επαγγελματική κατάρτιση σε άτομα τα οποία έχουν ε, σπουδάσει, έχουν ολοκληρώσει την, την εκπαίδευσή τους, να μεταβούν σε ένα κράτος μέλος άλλο και σε ένα καθεστώς ανταλλαγής να κατανοήσουν καλύτερα πού βρίσκονται και τι έχουν να κάνουν, αλλά να τους δώσουν και έμπνευση, με νέες προσεγγίσεις ε, ως προς την επιχειρηματικότητα. Αυτό θεωρώ ότι θα αποτελέσει μία από τις μεγάλες αλλαγές του μελλοντικού προγράμματος Erasmus Plus και τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία ήδη τώρα. Α, αλλά και στο μέλλον υπάρχει σχετική δέσμευση για επιπλέον χρηματοδότηση για άτομα τα οποία προέρχονται από μειονεκτικό υπόβαθρο γιατί το πρόγραμμα Erasmus δεν είναι επαρκές για να τα βγάλει κανείς πέρα στο πρόγραμμα αυτό, στο εξάμεινο αυτό αυτό. Και έτσι λοιπόν ε, δίδονται υποτροφίες σε άτομα τα οποία κάνουν ανταλλαγή στα πλαίσια του Εράσμους για να βοηθηθούν οι οικογένειές τους και αυτό θα ενισχυθεί και στη μελλοντική προγραμματική περίοδο. Για να υποστρεχθεί λοιπόν η προσπάθεια επαγγελματική κατάρτιση και αναβάθμιση των προσόντων των ατόμων αυτών στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Η κυρία Μωράν Σαρτιέ. Και μετά η κυρία Μακιντάε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ήταν εξαιρετική η παρουσίαση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλων των υφιστάμενων προγραμμάτων, όπω συνήθω. Και χαίρομαι ιδιαίτερω που ακούσα το πρόγραμμά σα για το θέμα αυτό τη ανάπτυξη τη μαθητεία με επιλογή των ε, μαθητευομένων σε ό,τι αφορά τον τομέα που θα ακολουθήσουν. Αλλά θεωρώ ότι σε ένα τομέα θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε μια προσπάθεια παραπάνω. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ε, της εξοικείωσης με τα σημερινά επαγγέλματα, γιατί συχνά τη βλέπουμε σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό της μαθητείας. Βλέπουμε ότι προσπούνται πολλοί ε, επαγγέλματα τα οποία είναι παροχημένα, επαγγέλματα τα οποία υπήρχαν, αλλά υπήρχαν ε, στην προηγούμενη γενιά ενδεχομένως. Αυτό που θα πρέπει να δείξουμε στους νέους, προκειμένου να τους παρακινήσουμε να στραφούν προς ένα επάγγελμα, είναι τι επαγγέλματα υπάρχουν ε, σήμερα. Και έχουμε μεγάλο έργο να κάνουμε στον τομέα της επικοινωνίας για να καταστήσουμε αυτά τα επαγγέλματα πιο ελκυστικά. Πώς έχουν εξελιχθεί λοιπόν τα επαγγέλματα σήμερα. Έχουν ε, εξελιχθεί πολύ. Αυτό πάντα συμβαίνει άλλωστε και θα πρέπει να τους δείξουμε πως έχει τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασία. Εδώ λοιπόν αντίθεται θέμα κουλτούρας, νοτροπίας που θα πρέπει να προωθήσουμε για να καταστεί πιο ελκυστική η μαθητεία. Και νομίζω ότι αυτό πραγματικά θα υποστηρίξει τους στόχους που έχετε θέσει και εσείς στο πρόγραμμά σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάκιντάιρ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να φτιάξουμε μεγαλύτερη σύνδεση των επιχειρήσεων και των ε, σχολών. Ένα πρόγραμμα σύντομων ε, πρακτικών ή μια σύντομη ε, εργασιακή εμπειρία είναι πραγματικά κάτι που λείπει. Ποιο το οργανώνει αυτά, δεν είμαι βέβαιη. Ίσως θα θέλετε να σχολιάσετε αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οργανώσεις όπως τα εμπορικά επιμελητήρια προκειμένου να διαμορφώσουν τον τρόπο παροχής ε, επαγγελματικής ε, κατάρτισης και να καλέσουν τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα εμπορικά μετρώα να δώσουν τέτοιες ε, δυνατότητες. Σε κάποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις μας λένε ότι δεν είναι πρακτικό ότι είναι επικίνδυνο, αλλά υπό κανονικέ συνθήκε όποιο ψάχνει βρίσκει ευκαιρίες. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Και ε, κυρίω για να υποστηρίξω αυτό που είπε η κυρία Μωράν Σορτιέ, ότι αλλάζει το εργασιακό περιβάλλον. Ο κόσμο ε, μπορεί να έχει κάποιε ιδέε ε, στο κεφάλι του, αλλά συχνά δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των μαθημάτων που παρακολουθεί κανεί στο σχολείο. Αγγλικά, μαθηματικά, γλώσσα και το καθεξής και των προσόντων που χρειάζεται στην αγορά εργασία τελικά. Και είναι δύσκολο ένας νέος να ξέρει τι πρέπει να μελετήσει στο σχολείο για να έχει μια επιτυχή καριέρα στη συνέχεια. Αυτό θα πρέπει να καταστεί πιο εύκολο ως μετάβαση για τους νέους, να γνωρίζουν καλύτερα τι χρειάζονται. Η ιδέα λοιπόν να υπάρχουν τέτοιες πιο πολλές ευκαιρίες για μαθητεία είναι αξιόλογη και αξίζει τον κόπο να δούμε τις πρακτικές δυσκολίες και τα πρακτικά, τις πρακτικές πτυχές της υλοποίησης αυτής της ιδέας, γιατί αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και τους βουλευτές και τους ε, προσκεκλημένους μας να σας ενημερώσω ότι οι συζητήσεις αυτές και οι εισαγωγέ, σα, οι παρεμβάσεις σας, συγγνώμη, ε, δημοσιεύθηκαν και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ακολούθησαν και σας παρακολούθησαν ε, πιο πολύ από όσοι βρίσκονται στην αίθουσα αυτή και άκουσαν τις προτάσεις σας και τη συζήτησή σας με τους ευρωβουλευτές. Ελπίζουμε δε να ξεκινήσουμε έτσι μια νέα παράδοση, την οποία και να επαναλάβουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. που απαντήσατε τα ερωτήματά μας και που παρουσιάσατε και τις δικές σας ιστορίες, τις δικές σας αξίες, τις δικές σας εικόνες όπως τις έχετε προσλάβει για το πώς θα μπορούσε δημορφωθεί ενδεχομένως στο μέλλον ή, εν πάση περιπτώσει, πώς θέλετε να διαμορφώσετε εσείς στο μέλλον. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εν παση περιπτωσει πως θελετε να δημορφώσετε εσεις συζήτηση και σας ευχαριστώ που ήλθατε και που αφιέρωσατε χρόνο για να μας παρουσιάσετε με μεγάλη λεπτομέρεια το τι κάνατε και τι ονειρεύεστε. Σας ευχαριστώ. Και θα συνεχίσουμε με το, υπό... με το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης ε, που αφορά μια παρουσίαση της μελέτης του Οργανισμού Θεμελιδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη αφορά την καταπολέμηση της παιδικής ε, φτώχειας ένα ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων. ανάμεσά μας είναι ο κύριος ε, ε, Γρηγόριος Τσιούκας, ο οποίος ε, ασχολείται με τα συγκεκριμένα ζητήματα στον Οργανισμό Θεμελιώδων Δικαιωμάτων. Θα παρουσιάσετε τη συγκεκριμένη μελέτη. Ξεκινάτε με έναν τίτλο αρχικά και στη συνέχεια. Περνάτε σε λεπτομέρειες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, πρόσκληση, ευχαριστώ την Επιτροπή σας ε, και τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την μελέτη μας ε, σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, ένα ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο τίτλος της μελέτης και φυσικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επίσης για την υποστήριξη που ε, δείχνετε προς το έργο μας ως Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στην παρουσίασή μου λοιπόν θα αναφερθώ στον στόχο της συγκεκριμένη έκθεσης και τα βασικά της μηνύματα και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω μια γενική εικόνα του περιεχομένου επικεντρωνόμενο σε δεδομένα, το νομικό πλαίσιο δράσης ε, κατά της παιδικής ε, φτώχειας και τα νομοθετικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάρκεια διάθεσή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, με βάση τις τελευταίες αναλύσεις και ευρήματα θα τονίσω μερικά ε, από τα ευρήματα των γνωμοδοτήσεών μας. Αυτή εδώ είναι η μελέτη για όσους ε, δεν το γνωρίζουν. Θα την ε, βρείτε και στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα μας. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στις 17 Οκτωβρίου, η Παγκόσμια ημέρα κατά της φτώχειας και αποτελεί επίσης και έναν χρόνο περίπου μετά την διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε ε, το, ε, πώς, ε, το σχεδιάγραμμα της παρουσίασής μου στόχους, βασικά μηνύματα, δεδομένα, κάποια λόγια για το νομικό πλαίσιο, τα ε, εργαλεία πολιτικής ε, και οι απόψεις μας. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν διότι ήδη είναι περασμένη ώρα και φαντάζομαι είστε όλοι κουρασμένοι. Ποιο λοιπόν είναι ο στόχος αυτής της μελέτης αρχικά να ενημερώσει ότι η παιδική φτώχεια είναι μια πραγματικότητα για μεγάλο αριθμό παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα πολύ σχετικό για την Ευρώπη και η Ευρώπη δεν εξαιρείται από το φαινόμενο της φτώχειας ε, η παιδική, και την παιδική φτώχεια ιδιαίτερος. Θα ήθελα να συνεισφέρω λοιπόν ε, σε αυτή την συζήτηση για μια πιο κοινωνική Ευρώπη, για τα δικαιώματα των παιδιών. Η γραμμή από την οποία ξεκινούμε είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινωνική Ευρώπη αν δεν κάνουμε αρχικά κάτι κατά της φτώχειας και συγκεκριμένα κατά της παιδικής φτώχειας. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ε, παιδική φτώχεια με περίπου 25 εκατομμύρια παιδιά τα οποία βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Ένα λοιπόν από τα βασικά μας μηνύματα είναι ότι θέλουμε να ε, τονίσουμε ότι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας δεν είναι μονάχα ένα ζήτημα επιλογών πολιτικής ε, και προτεραιοτήτων αποτελεί επίσης ένα ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων, το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα ζήτημα νομικά δεσμευτικών ε, ε, υποχρεώσεων τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τα κράτη-μέλη αλλά και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς διότι πολλά παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να πληρώσουν ε, για βασικά πράγματα όπως είναι διακοπές, αυτοκίνητα, υπολογιστές. Αυτό είναι πολύ ενισχυτικό. Από την άλλη όμως ε, το να ε, μην να στερείς τα πιο βασικά όπως είναι οι εγκαταστάσεις Ε, Υγεία ε, ηλεκτρισμού, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ε, θέματα και είναι κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τι δείχνουν λοιπόν τα δεδομένα. Έχουμε περίπου 25 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο σημαίνει ένα στα τέσσερα παιδιά τα οποία ε, ζουν ε, υπό κίνδυνο φτώχειος ή κοινωνικού αποκλεισμού. Περίπου 2 εκατομμύρια από αυτά αντιμετωπίζουν ε, και τις τρεις εκφάνσεις της φτώχειας, το οποίο σημαίνει ότι ζουν κάτω από το ε, όριο της ε, εισοδηματικής φτώχειας, όπως ορίζεται από την Eurostat, ε, αντιμετωπίζουν σημαντικές θερήσεις και ταυτόχρονα ζουν σε νοικοκυριά όπου υπάρχει ελάχιστη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ισχύει ότι η τάση τα τελευταία χρόνια δείχνει ε, μία μείωση ε, στον αριθμό των παιδιών ε, που ζουν σε καθεστώς στάχια σε σχέση με το 2012. Βλέπουμε ότι το ποσοστό για το 2012 ήταν στο 28% ενώ η τελευταία, τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, ε, αν θυμάμαι πέρσι το Σεπτέμβρη, ε, δείχνουν μία πτώση της τάξης του 4%. Παρ' όλα αυτά όμως οι αριθμοί παραμένουν πολύ υψηλοί και ο αριθμός των παιδιών που ζουν σε καθεστώς φτώχειας είναι υψηλότερος από τους αριθμούς που αφορούν τον γενικότερο πληθυσμό. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι τα παιδιά είναι αυτά τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από την φτώχεια σε σχέση με τους ε, ανθρώπους άνω των 18. Ένα άλλο θέμα είναι ότι υπάρχει, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφορών κρατών μελών. Για παράδειγμα, ε, Βουλγαρία, Ρουμανία το 40% και πάνω των παιδιών ε, ζει υπό κίνδυνο φτώχειος ενώ σε Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Ισπανία το ποσοστό αυτό είναι στο 30% ορισμένες ε, ομάδες παιδιών όπως τα παιδιά Ρωμά ή παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο αντιμετωπίζουν ε, πολύ χειρότερες ε, συνθήκες. Άλλοι παράγοντες ε, είναι επίσης το πώς είναι το νοικοκυριό τους. Για παράδειγμα, μονογονεϊκές οικογένειες ή μεγάλες οικογένειες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα όπως επίσης και το χαμηλό εκπαιδευτικό ε, υπόβαθρο των γονέων. Όσο πιο χαμηλό είναι το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο των γονέων, ε, τόσο υψηλότερο ε, είναι ο κίνδυνος φτώχειας για τα παιδιά. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε ένα χάρτη ο οποίος παρουσιάζει τα ευρήματά μας. Βλέπετε λοιπόν σε Ποιε χώρες είναι η κατάσταση πιο σοβαρή, αυτά τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Ποιε χώρε λοιπόν έχουν ε, υψηλότερα ποσοστά και ποιε ε, είναι σε καλύτερη κατάσταση, να το θέσουμε έτσι. Αυτός ο πίνακας τώρα, αυτό το διάγραμμα τώρα, σας κάνει μια σύγκριση μεταξύ ε, παιδιών του γενικού πληθυσμού και παιδιών ε, Ρωμά και μπορείτε ε, να δείτε ότι πρόκειται για δεδομένα τα οποία προέρχονται από δική μας έρευνα του οργανισμού και της EU Mindis που έγινε το 2016 και όπου μετρήσαμε μεταξύ άλλων την ε, φτώχεια ε, και το πώς βιώνεται σε νοικοκυριά Ρωμά και ε, νοικοκυριά μεταναστών. Εδώ βλέπετε τα νοικοκυριά Ρωμά και μπορείτε να δείτε ότι σε ότι οι αριθμοί ε, κάνουν τρομερή εντύπωση. Πάνω από το 90% των οικογενειών ε, Ρωμά, σύμφωνα με ε, τις απαντήσεις στην έρευνά μας, αντιμετωπίζουν συνθήκες φτώχειας. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα. Τώρα ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. η καταπολέμηση της ε, παιδικής φτώχειας είναι και ε, νομική υποχρέωση, δεν αποτελεί μονάχα ε, πολιτική προτεραιότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 24 της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ανθρωπίνων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων διασφαλίζει το την προστασία των παιδιών και την διασφάλιση της ευημερία τους. Επίσης έχει νομική αξία διότι ε, υπάρχει στις συνθήκες το οποίο σημαίνει ότι είναι δεσμευτική για τους ε, θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε την ευρύτερη εικόνα σε διεθνές επίπεδο όλα τα κράτη-μέλη, και πιθανότατα αυτή είναι μία από τις λίγες ε, συμβάσεις του ΙΕ που έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του ΙΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου έχουμε έναν ευρύ κατάλογο δικαιωμάτων που αφορούν τα παιδιά, κυρίως ε, σε ό,τι αφορά ε, δικαιώματα που αφορούν την καταπολέμηση της παιδικής ανέχειας. Ε, Παίρνοντα χάρη στη σύμβαση αναγράφεται το δικαίωμα κάθε παιδιού σε ένα επαρκές βιωτικό επίπεδο, άρθρο 27. Και επίσης όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, νομικές υποχρεώσεις ε, σε σχέση με οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα στο πλαίσιο του συστήματος ε, συνθήκων της, ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βεβαίως δεν δεσμεύονται όλα τα κράτη-μέλη από τις ίδιες διατάξεις ε, του χάρτη και δεν έχουν επικυρώσει ή έχουν θετήσει όλα τα κράτη-μέλη τον θεωρημένο κοινωνικό χάρτη. Όμως, Ο χάρτης αποτελεί όχι μόνο πηγή έμπνευση για τη δουλειά μας, αλλά πολλές από τις διατάξεις του, το χάρη το άρθρο 17, προβλέπει την προστασία των παιδιών και των οικογενειών. another ε, ε, issue regarding ε, the legal framework, let's say, it is true that... Ένα άλλο θέμα που αφορά το νομικό πλαίσιο. Είναι αλήθεια ότι καταρχήν η αρμοδιότητα έγκυται στα κράτη-μέλη. Επομένως, η δουλειά που πρέπει να κάνουν οι εθνικές αρχές είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ σημαντικές αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά την υποστήριξη που πρέπει να δώσει στα κράτη-μέλη για να συμπληρωθούν οι προσπαθίες τους. Τώρα, τα εργαλεία πολιτικής. Ε, μιλήσαμε για τα απορίσματα, μιλήσαμε για το νομικό πλαίσιο, πώς απαντάμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Έχουμε τη σύσταση του 2013, επενδύοντας τα παιδιά που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι φυσικά ένα μέσο μη δεσμευτικής νομοθεσίας, αλλά δίνει απάντηση νομοθετικής ό,τι αφορά την ανέχεια των παιδιών. Έχουμε τρεις πυλώνες. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι γονείς έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πόρους, είτε μέσω της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, είτε μέσω επαρκών ε, κοινωνικών επιδομάτων. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας. Ε, ο δεύτερος πυλώνας αφορά την πρόσβαση των γονέων και των παιδιών σε ε, ποιοτικές και φθηνές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στη στέγαση και σε εναλλακτικέ δομές φροντίδας ε, και τρίτον η πρόθεση του δικαιώματος των παιδιών να συμμετέχουν και στην ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ε, σήμερα το πρωί είχαμε μία εκδήλωση στο ίδιο κτίριο, γιατί σήμερα είναι, γιορτάζουμε την επέτειο των δικαιωμάτων των παιδιών και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που οργανώθηκε για τα δικαιώματα του παιδιού και ακριβώς αναφέρθηκε το θέμα της ε, συμμετοχής εκτενώς. There were some quite ε, promising uh, results coming. Και υπάρχουν κάποια υποσχόμενα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μελέτη που υλοποιήθηκε από το Eurochild. Προχωρώντας, η έκθεση δεν αναλύει απλώς το πλαίσιο πολιτικής και τα γεγονότα, αλλά αναφέρεται και σε συγκεκριμένα εργαλεία πολιτικής που έχουμε στη διάθεσή μας. Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Ξάμεινο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν λαμβάνει επαρκώ υπόψη το θέμα του δικαιωμάτων του παιδιού και τη ε, παιδική ανέχεια. Οι ειδικέ συστάσει αναχώρα που σχετίζονται με τα παιδιά συνήθω αναφέρονται σε υπηρεσίε φροντίδα, ε, στην εκπαίδευση ή στην ε, εκπαίδευση σε σχέση με την ένταξη. Παρ' όλα αυτά, αναφορέ ε, στην παιδική φτώχεια ω τέτοιε λείπουν. Το 2018, παραδείγματο χάρη, μόνο μία δική σύσταση ανά χώρα ρητά ε, στόχευε στην παιδική φτώχεια. Ένα άλλο πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Στην έκθεσή μας προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις προτάσεις της Κομισιόν σε ό,τι αφορά το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εδώ τα πήσαμε κάποια ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία. Παραδείγματο χάρη, μια πιο κοινωνική Ευρώπη που εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων είναι μεταξύ των γενικών στόχων πολιτικής και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και για το ΕΤΠΑ. Η ε, συγκεκριμένοι στόχοι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΕΙΝ ε, και τη σχετική χρηματοδότηση αναφέρονται ρητά στα παιδιά ως ε, πιθανή δικαιούχοι δράσεων ενώ το σχέδιο του νέου κανονισμού περί κοινών διατάξεων προτείνει να συμπεριληφθούν σκέψεις περί παιδικής στόχιας στο νέο σύστημα αιρεσιμότητας που προτείνεται για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι τα γνωρίζετε όλα αυτά. Επίσης, αναφέραμε την, το δυναμικό του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε αυτό το πλαίσιο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ ιδιωτική και επαγγελματική ζωή, γιατί αυτό προωθεί τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και έτσι συμμετέχουν στην καταπολέμηση παιδικής φτώχειας. Επίσης, ε, ο κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων είναι ένα σημαντικό θέμα. Μετρά την πρόοδο στην εφαρμογή του πυλώνα και φυσικά η εγγύηση για τα παιδιά που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να πετύχουμε ότι κάθε παιδί σε κατάσταση ανέχειας μπορεί να έχει πρόσβαση σε δωρεάν περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή τροφή. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υλοποιείται μια μελέτη σκοπιμότητας για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με την αγγίση για τα παιδιά. Και τέλος, η έκθεσή μας περιλαμβάνει μία σειρά συγκεκριμένων απόψεων για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Αφορούν πέντε τομείς, καταρχήν. Νομοδοτήσεις για το πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε το νομικό πλαίσιο, να ενισχύσουμε το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση παιδικής φτώχειας. Πώς θα ευθυγραμμίσουμε την ευρωπαϊκή δράση με τα νομικά πρότυπα που συμπεριλαμβάνονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Παιδιών αλλά και τον Ευρωπαϊκό, Χάρτη Κοινωνικών τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και επίσης πώς θα γίνει η προσχώρηση στον εθεωρημένο κοινωνικό χάρτη από τα κράτη-μέλη. Εξετάζουμε και πώς θα προωθήσουμε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Το δεύτερο αφορά την επικέντρωση στους πιο ευπαθείς ομάδες, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει κινδύνος παραβίασης των δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η θέσπιση της εγγύησης για τα παιδιά μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος, για να αντιμετωπίσουμε την οξία ανέχεια και θεωρούμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα την προστασία των παιδιών σε ευάλωτες καταστάσεις, κυρίως τα παιδιά Ρωμά και κυρίως ε, παιδιά με υπόβαθρο μεταναστευτικό, παιδιά με αναπηρίες, ε, παιδιά που ζουν σε μεγάλες οικογένειες ε, ή σε μονογονεϊκές οικογένειες. Το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς πολιτικής να προστατεύσουμε τα παιδιά από την ανέχεια. Θα πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου τη σύσταση του 2013, κυρίως ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και θεωρούμε ότι οι ειδικέ συστάσεις αναχώρας, αναχώρας συγγνώμη, θα ήταν χρήσιμο να προσανατολίζονται περισσότερο στα παιδιά. Ένας άλλος τομέας είναι αυτό που αποκαλούμε ανάληψη δράσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ήδη ανέφερα την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ ιδιωτική και επαγγελματική ζωής. Επίσης χρήσιμο θα είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων για να εγκατοπτρίζεται και η κατάσταση των παιδιών. Έχουμε δεδομένα, η Eurostat μπορεί να παρέχει πολλά δεδομένα. Ο πίνακας αποτελεσμάτων σε σχέση με τα παιδιά. Μπορεί να μας δώσει αναλυτικά δεδομένα για τα παιδιά. Θα μπορούσε λοιπόν να αντικατοπτρίζεται να αντικατοπτρίζονται αυτά τα αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα αποτελεσμάτων. Και τελευταίος ε, τομέας αφορά την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ε, καταπολέμησης της παιδικής στόχιας, γιατί χωρίς την κατάλληλη χρηματοδότηση τα διάφορα σχέδια και προγράμματα δεν μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα. Uh, Θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά που ζουν σε κατάσταση φτώχειας ή σε κατάσταση αποκλεισμού αποτελούν ε, προτεραιότητα υπό το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, όχι μόνο ε, προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αλλά και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε αυτό που αποκαλούμε κατάλληλες προϋποθέσεις, enabling conditions για την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση συμπεριλαμβανούν και σκέψεις και προβληματισμούς που αφορούν τα παιδιά. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you uh, for your... Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει Πρόεδρος, για την ε, εξαντλατική και ιδιαίτερα λυπηρή αυτή η απεικόνηση της πραγματικότητας. Ε, δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις, κυρία Λάμπερτ, έχουμε πέντε λεπτά μόνο, γι' αυτό θα πρέπει να βιαστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η παρουσίαση πρόσφατα. Ενημερώθηκα για τη δήλωση του δικού επιστολμένου του, τον είπα για τα θέματα φτώχειας μετά από επίσκεψη του στο Ενωμένο Βασίλειο. Και αυτό είναι ακόμα πιο καταθλιπτικό. Ένα από τα θέματα που έθιξε για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τα διάφορα μέτρα τα οποία χρησιμοποιεί το Ενωμένο Βασίλειο που σημαίνει ότι μπορεί να προσαρμόσει κανείς τις απαντήσεις του στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Θα ήθελα να μας πείτε, έχετε σχόλια να κάνετε από την έρευνά σας ε, για το πώς μετράτε η φτώχεια. Είμαστε συνεπείς στην μέτρηση των στοιχείων αυτών και των δικτών. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι από το εξή. Λαμβάνουμε υπόψη τα στοιχεία τα οποία μας χορηγεί η Eurostat. Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία αυτά που μας δίνει η Eurostat. Είναι η γραμμή φτώχειας, το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος. Τα άτομα που είναι κάτω από το επίπεδο λοιπόν αυτό. Αλλά δεν μόνο το θέμα της φτώχειας σε ό,τι το εισόδημα. Δεν μετρά μόνο αυτό. Τίθεται και το θέμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως προκύπτει από την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Η Eurostat λοιπόν χρησιμοποιεί τον δίκτυ της υλικής των υλικών ελλείψεων και αυτό έχει να κάνει με πρόσβαση σε νέα διαφορετικά προϊόντα, αγαθά. Για παράδειγμα, το κατά πόσο ένα νοικοκυριό μπορεί να πληρώσει τον οίκαιο του τους λογαριασμούς του, ε, το αυτοκίνητο, το τηλέφωνο, τις διακοπές. Υπάρχει λοιπόν ένας κατάλογος με νέα τέτοια διαφορετικά στοιχεία και σοβαρή έλλειψη τέτοια ελική έλλειψη αγαθών και υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι φύσταται όταν δεν μπορεί κανείς να έχει χρήματα για τέσσερις από τις εννέα αυτές κατηγορίες. και το θέμα της ανεργίας σε επίπεδο νοικοκυριού. Έχουν οι γονείς, για παράδειγμα, πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Έχουν πλήρη απασχόληση, μερική απασχόληση, τι είδου απασχόληση. Όλα αυτά παίζουν ρόλο για να προσμερτηθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, γιατί προφανώς πρόκειται για δείκτες. Η φτώχεια αποτελεί δείκτη, κοινωνικό αποκλεισμό αποτελεί δίκτυ Και ένα σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι το εξή. Η Eurostat και οι Εθνικέ Στατιστικέ Υπηρεσίε δεν λαμβάνουν υπόψη και κάποια εθνοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού σε ό,τι αφορά τους Ρωμά. Στην πράξη είναι δύσκολο να προσμετρηθεί η φτώχεια. Σε ό,τι αφορά τμήματα του πληθυσμού, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερε δυσκολίε. Όχι μόνο οι Ρωμά, αλλά και άτομα από πρόσφυγες, ε, άτομα με αναπηρία. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε ήταν πραγματικά καταθλιπτικά. Μιλάμε για 25 εκατομμύρια παιδιών στο πιο πλούσιο κομμάτι του κόσμου. 25 εκατομμύρια παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Καταστροφικό. Ελπίζω να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα και στους κόλπους της Επιτροπής μας και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ότι αυτό είναι ένα θέμα της καθημερινής ζωής ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά παιδιά, γιατί υπάρχει τάση να το ξεχνάμε αυτό. Ελπίζω λοιπόν και εσείς να το φροντίσετε αυτό, προκειμένου να περάσει αυτό το μήνυμα σε όσους πιο πολύ γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο. Προκειμένου να ενημερωθούν τουλάχιστον όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα γεγονότα. Είναι δημόσια τα στοιχεία αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας μέχρι τέλους στη συνεδρίαση της, ομα... της Επιτροπής μας. Επόμενη συνεδρίαση στις 27 Νοεμβρίου εδώ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ.